Okay, uh, we start the meeting and... Uh, λοιπόν, φίλοι μου, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε όλοι, πρόκειται για νέα θητεία και έχουμε διορισμό νέων μελών στην Επιτροπή και γι' αυτό το λόγο και για άλλους λόγους έχουμε καλέσει τους διευθυντές των τεσσάρων οργανισμών που ασχολούνται με θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για μας στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θέλουμε λοιπόν να τους ακούσουμε, να ακούσουμε με τι ασχολούνται αυτοί ακριβώς στη στιγμή, τι έχουν κάνει προηγουμένως και τι σκοπεύουν να επιτύχουν με την εργασία τους, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση των οργανισμών αρχίσουμε με τον κύριο James ε, Καλέχα, που είναι Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ΣΕΔΕΦΟΠ, όπως είναι γνωστό περισσότερο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις υπόλοιπες εισηγήσεις και μετά έχουμε μια περίοδο ερωταπαντήσεων. Κύριε Καλέχα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτέ, Καταρχήν να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι όχι μόνο χαρά αλλά και προνόμιο να είμαι σήμερα εδώ. Είναι μια από τι συνεδριάσει όπου εγώ αισθάνομαι πιο κοντά στου ευρωπαίου πολίτε, διότι εσεί αντιπροσωπεύετε του Ευρωπαίου πολίτε εδώ και εμεί εργαζόμαστε για του Ευρωπαίου πολίτε. Πραγματικά λοιπόν μεγάλη μου τιμή και να μιλήσω για αυτό το κέντρο που είναι ένα οργανισμό που καλύπτει όχι μόνο την απασχόληση αλλά και την απασχόληση απασχολησιμότητα και ποικίλει ανάμεσα στο σχολείο μέχρι την ε, ηλικία της συνταξιοδότησης. Είναι μια από, ένας από τους παλιότερους οργανισμούς, ε, ιδρύθηκε το 1975. Περάσαμε 20 χρόνια στο Βερολίνο και μετά ο οργανισμός μας μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ε, Έχουμε ε, προπολογισμό 80 εκατομμύρια ε, και προσωπικό 23 ατόμων. Δημιουργήθηκε ο οργανισμός μας μέσω του κανονισμού 337 του Συμβουλίου. Εμείς Στοχεύουμε στην υψηλή ποιότητα επαγγελματική κατάρτιση που είναι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και στην αγορά εργασίας. Αυτό το οποίο καλύπτουμε λοιπόν είναι η σχέση ανάμεσα στις δεξιότητες, τα προσόντα και την απασχολησιμότητα. Και έχουμε τρία ερωτήματα που πάντοτε ε, βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος εργασίας μας, δηλαδή το πώς θα συνδυάσουμε ένα υψηλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό με την κατάλληλη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πώς θα αυξήσουμε τη συμμετοχή σε μια συρρυκνούμενη και γυράσκουσα αγορά εργασίας και το τρίτο ερώτημα είναι πώς η κατάρτιση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την ε, ανισότητα και να προωθήσει την ε, πράσινη οικονομία interface, ε, αλληλεπίδραση δηλαδή ανάμεσα στην κατάρτιση και την αγορά εργασία. Εν γέννη έχουμε τρει προτεραιότητε από τον οποίο εστιάζουμε. Πρώτον, εξυγχρονισμό τη επαγγελματική κατάρτιση, η χειραφέτηση των ανθρώπων, των ατόμων στη σταδιοδρομία τους και η δυνατότητα μετάβασης σε μια, ένα μεταγενέστερο στάδιο της απασχόλησής τους, της σταδιοδρομίας τους και έπειτα αναλύουμε τις ε, δεξιότητες προβλέποντας τι θα χρειαστεί η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Το 2013 ε, το Συμβούλιο δήλωσε ότι η εργασία μας ως οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεγάλη, χέρι μεγάλη εκτίμηση και εκτός Ένωσης. Ε, είμαστε αναγνωρισμένοι ως ε, ένα κέντρο αριστείας όσον αφορά την, ε, τις ε, δεξιότητες και την ε, αντιστοιχεία αυτών με τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, όσον αφορά την απασχόληση και την απασχολησιμότητα, την κατάρτιση μάλλον και την απασχολησιμότητα και τέλος οι εξωτερικές αξιολογήσεις είπαν ότι δεν επικαλυπτόμεθα στην εργασία μας την εργασία άλλων οργανισμών της Ένωσης. Η εργασία μας λοιπόν χρησιμοποιείται ευρύτατα. Για να σας δώσω κάποιες ιδέες, από το 2005 είχαμε 96,6 εκατομμύρια επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Είχαμε 42 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι κατέβασαν και χρησιμοποίησαν το, το Γεωγραφικό σημείωμα Europass. Ε, πέρυσι είχαμε 173 παραπομπές σε ευρωπαϊκά έγγραφα. Πρόκειται για αύξηση 12% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το 2013 πάνω από 6.036 ε, ε, μάλλον 636.000 δημοσιεύσεις έγιναν και ε, αναγνώστησαν από τους Ευρωπαίους πολίτες για να, ένα δείγμα για το πόσο πολύ έχει χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπός μας τα τελευταία χρόνια. Τώρα, εφόσον έχουμε δυνατότητα πρόσβασης ε, στην έρευνα, είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό που είναι και εξίσου σημαντικό είναι το μήνυμα που διαβιβάζει ο οργανισμός του Σεντεφόπ στα κρατημέλη. Και το μήνυμα αυτό είναι σαφές ότι χρειάζεται επαγγελματική κατάρτιση που να είναι ελκυστική, να είναι για όλους, να είναι προσιτή και ευέλικτη. Υπάρχει μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2002, την οποία παρακολουθήσαμε στενά με την ε, Επιτροπή και πρόκειται για την ε, διαδικασία της Κοπεχάγης που τελειοποιήθηκε με το ανακοινοθέν του 2010. Θέλουμε να μεριώσουμε τους ε, εγκαταλείποντες πρόεδρες στο σχολείο και θέλουμε να θαρρύνουμε τον κόσμο να μείνει στη διαβίου ε, μάθηση. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, να συγκεντρώσουμε κοινωνικούς εταίρους κράτη-μέλη, ώστε από κοινού να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο κείμενο επί το οποίο συμφώνησαν οι Υπουργοί Παιδείας ε, το 2010. Πρόκειται για το ανακοινωθέν της Ε, αν εσείς, ε, τα κράτη-μέλη, ε, τα, το, εσείς οι προβουλευτές ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τον ανακοινωθέν της Μπρούζη, αλλά και να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία μέσα, ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν την ε, ενέργεια και την διαδικασία μεταρρύθμισης που χρειάζεται στην, στην, κλιματική κατάρτιση, όπως ας πούμε, το πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά προσόντα, η το ίσω το οποίο να έχετε συναντήσει, το Europass που σα ανέφερα πριν από λίγο, ή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίηση για την Επαγγελματική Κατάρτιση, ή την επικύρωση τη μη επίσημη ή άτυπης ε, ε, μάθησης. Ε. Όλα αυτά είναι συστάσεις που το Ευρωκοινοβούλιο έχει συμφωνήσει στη διάρκεια των ετών. Τώρα, σε ποιο βαθμό έχουν χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια των ετών, έχουν χρησιμοποιηθεί και πολλές χώρες τα χρησιμοποιούν και σήμερα αυτά τα μέσα. Αλλά η έκκλησή μου προς εσάς είναι να ενθαρρύνετε περισσότερο τα κράτη-μέλη σας να χρησιμοποιούν αυτά τα ευρωπαϊκά μέσα. Πρόκειται και ευρωπαϊκά μέσα, επαναλαμβάνω, που δίνουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, δεξιότητες και στα πτυχία αυξάνουν την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, δίνουν περισσότερη προσβασιμότητα στην ε, επαγγελματική κατάρτιση και ελκυστικότητα και επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες να είναι ε, ε, ευκίνητοι εσωτερικά αλλά και μέσα, ανάμεσα στα κρατημέλη. Ένας άλλος τομέας ανάλυσης είναι βέβαια το τι κάνουμε για τις μεταβατικές μάλλον για τη μετάβαση στη διάρκεια μιας αδιαδρομίας. και αυτό είναι δηλαδή το θέμα της διαβίου μάθησης. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να παραμείνουν απασχολήσιμοι. Δεν είναι μόνο η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη ώστε να μπουν σε τομείς όπως προγράμματα μαθητείας ή μάθηση μέσω του δικτύου θα ξεκινήσουμε τώρα ένα νέο πρόγραμμα για το κόστος και τα ωφέλη ενώ, ε, ε, τέτοιων ε, προγραμμάτων για τα κράτη-μέλη. Ένα από τα διδάγματα που πήρα όταν, όσο έζησα στην Ελβετία ήταν ότι όσο περισσότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταρτίζουν τους υπαλλήλους τους, τόσο περισσότερα ωφέλη αποκομίζουν. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που πιστεύω οι εταιρείε μας θα πρέπει να το πάρουν πολύ σοβαρά. Τώρα, όταν κανείς έρχεται ως θεσμός στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ, η δική μου πρόσκληση προς εσάς είναι ε, ότι πρέπει να ε, ε, να συνδυάσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας. Ε, ο οργανισμός είναι ένας ευρωπαϊκός ανεξάρτητος πόρος, αλλά πέρα από αυτό εγώ θα ήθελα να δω στους οργανισμούς της Ένωσης να ε, γίνονται πιο σχετικοί με τις δικές σας εργασίες, τους οδικούς χάρτες, τις δικές σας ιδέες για τα επόμενα χρόνια Ναι, γιατί έτσι νομίζω θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό μας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Πέρυσι φτάσαμε στο 99,5% όσον αφορά την απορρόφηση του προπολογισμού μας, αλλά θέλουμε περισσότερη επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο και τα κρατημέλη, γιατί μόνο όταν κανείς αγγίζει τη βάση της κοινωνίας, συνειδητοποιείς πόση δουλειά πρέπει να γίνει και τι δουλειά πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των πολιτών μας. Είμαστε λοιπόν ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που θέλει να μετατρέψει τις αδυναμίες σε δύναμη ε, και τα ισχυρά σημεία σε βιωσιμότητα. Έχουμε διάφορα πρότυπα για το πώς η επαγγελματική κατάρτιση έχει μετατρέψει τις οικονομίες μεταμορφώσει της οικονομίες εκεί όπου η επαγγελματική κατάρτιση είναι ισχυρή, η ανεργία ιδιαίτερα των νέων είναι πολύ χαμηλή, ενώ το αντίστροφο επίσης συμβαίνει θέλουμε να εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε την ε, ε, συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ε, πληροφορίες για να εντοπίσουμε κοινέ ευρωπαϊκές προσεγγίσεις και αρχές για να βελτιωθεί αυτή η σχέση και εξυπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε ε, να χρησιμεύουμε μάλλον ως σημείο συνάντησης για τους ηθήνοντες της χάραξης της πολιτικής. Φυσικά παραμένουμε ένας Ευρωπαίος ε, το βασικό μας στόχος είναι ο Ευρωπαίος πολίτης, ε, ο άνθρωπος που έχει από στην κοινωνία γιατί δεν έχει δουλειά. Εκεί είναι η αιστεία μας και η προτεραιότητά μας και θα κλείσω λέγοντας ότι έχουμε αφήσει εδώ έξω από την αίθουσα υλικό, κοιτάξτε να χρησιμοποιήσετε τους σπόρους μας και ελάτε σε επαφή μαζί μας όποτε αν χρειαστείτε πληροφορίες ή αν χρειαστείτε κάποιες λεπτομέρειες για την δουλειά σας, μπορεί να σε βρεθεί στη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χουάν Μενέντες Βαλντές, που είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, το Eurofound, που τον είδατε και προηγουμένως νωρίτερα, όταν συμμετείχε στην συζήτηση για την αδήλωτη εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαστε ένας οργανισμός με πολύ μεγάλο όνομα. Η σύντομη εκδοχή είναι Eurofound και θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την ικανοποίησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ε, δύο λόγια με αυτά που βλέπετε εδώ στην οθόνη, αν μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες. Μπορεί να είστε εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους, γιατί αυτά είναι τα θέματα τα οποία ε, σας απασχολούν περισσότερο και αυτά που χρησιμοποιείται πιο συχνά όταν έρχονται επίτροπε και αντιπρόεδροι εδώ ε, για τον κοινωνικό διάλογο, για την ε, ε, θέση απασχόλησης, για την ανάπτυξη. Και ήθελα να τις επισημάνω αυτές τις λέξεις, διότι όλοι αυτοί οι όροι είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας έρευνας και επικοινωνία στο Eurofound και θα ήθελα να ξεκινήσω την παρουσίασή μου με κάποια παραδείγματα από τις διαπιστώσεις μας από τις έρευνες αυτές, ε, που είναι στο επίκεντρο αυτών που σας αποσχολούν, που, εδώ στο, που συζητάτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα των θέσεων εργασίας και των διαθροτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας. Αυτά τα παρακολουθούμε μέσω του European Jobs Monitor που ε, ε, βλέπουμε ε, τα καθαρά κέρδη και τις καθαρές απώλειες σε θέσεις εργασίας σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ή χάθηκαν στην Ευρώπη. Πρόκειται για εργασίες διαφόρων ειδών ε, και διαφορετικού μισθών Έχουμε δηλαδή ε, θέσεις ελάχιστο κατώτατων μισθών, αλλά ε, είδαμε ότι στη διάρκεια της ύφεση υπήρχαν ε, αυξήσεις και στις υψηλόμισθες ε, θέσεις εργασίας και στις χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας και κάνουμε μια σύγκριση και βλέπουμε τι γίνεται και με τους εργαζομένους και το 2015 θέλουμε να δούμε την πολλοπλικότητα των θέσεων εργασίας βάσει καθηκόντων. Ε, επίσης, έχουμε τον κοινωνικό διάλογο βεβαίως που σας αφορά και εσάς και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνάς μας. Είμαστε τριμερής ε, οργανισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσώπους των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων όπως ε, γίνεται και στις ΕΝΤΕΦΟΠ ε, και ε, και εμείς έχουμε μια σειρά από προγράμματα ερευνητικού χαρακτήρα ε, στη διάρκεια για παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Εξαμένου, τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας και τι γίνεται και στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που συζητάτε και εδώ. Και εξετάζουμε όχι μόνο τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου. Παραδείγματο χάρη, συλλογικέ συμβάσει, κατώτατε μισθή ή ε, χρόνο εργασία σε συλλογικέ συμβάσει. Ε, σε σχέση με αυτό έχουμε αρκετά προγράμματα τα τελευταία έτη, πώς έχουν επηρεάσει τους μισθούς και τον καθορισμό των μισθών και τον μηχανισμό καθορισμού, ε, τα μνημόνια ε, συνεννόησης για παράδειγμα στις χώρες τις οποίες έχουν μνημόνιο και καθώς επίσης και τις συλλογικές συμβάσεις με τους κατώτατους μισθούς ε, και ε, εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες και αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα για τις ανισότητες ε, στους μισθούς. Θα σας παρουσιάσουμε και κάποια προκαταρκτικά ευρήματα σε ένα γεύμα εργασίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Νοεμβρίου. Ε, ένα ακόμα θέμα το οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί ε, σχετίζεται με την αδήλωτη εργασία. Εδώ έχουμε μια βάση δεδομένων με μέτρα ε, καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Αυτό ήταν στα πλαίσια ενός προγράμματος για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Ένα άλλο που σας αφορά είναι η ποιότητα της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες. Γνωρίζουμε ότι βάση των στοιχείων της Eurofound και της έρευνας για, το για την ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών είναι ακόμα πιο σημαντική ε, από την αντίληψη της οικονομικής απόδοσης μιας χώρας και έχουμε αναπτύξει ε, μια σειρά από διάφορα ερευνητικά προγράμματα που εξετάζουν διάφορες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα υπηρεσίες ε, φροντίδας παιδιών και πώς εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές χωρίς ταυτόχρονα να υποσκάπτουν την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Υπάρχει και κάτι ακόμα ε, με το οποίο είστε εξοικειωμένοι. Εδώ έχουμε τους μακροχρόνια άνεργους, τους λεγόμενους νίτς, ε, ανθρώπους που ούτε είναι σε διαδικασία εκπαίδευσης, ούτε κατάρτισης, ούτε έχουν κάποια θέση εργασίας. Ε, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται με την ανεργία των νέων και κοιτάμε το κόστος της αδράνειας και εξετάζουμε και άλλες περιπτώσεις. Ε, το Eurofund λοιπόν ε, κάνει ε, αντίστοιχη εργασία. Ω προς τα μεγέθη μας είμαστε αντίστοιχοι με το ε, Εδρεύουμε στο Δουβλίνο, ε, ιδρυθήκαμε από το 1975, μαζί με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ είμαστε ο, οι αρχαιότεροι οργανισμοί, του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια μας και ε, είμαστε και στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανισμών στην Ευρώπη η αποστολή μας. όπως ε, αναφέρεται στο τετραετές πρόγραμμά μας, είναι πολύ απλή. Θέλουμε να παρέχουμε γνώση για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη κοινωνικών και ε, ε, πολιτικών εργασίας ε, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο ενημερωμένες πολιτικές. Προσπαθούμε λοιπόν να σας βοηθήσουμε και αυτό είναι και ο τίτλος του τετραετούς προγραμματός μας και εξετάζουμε τέσσερις διαφορετικούς τομείς, ένας ο οποίος σχετίζεται στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή της και την ανεργία, ένας δεύτερος στις εργασιακές συνθήκες, πώς μπορούν να είναι πιο βιώσιμες με βάση και τις δημογραφικές αλλαγές και την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και ο τρίτος σχετίζεται με τις βιομηχανικές Πώ σχέσεις, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοιες σχέσεις, τέταρτος ε, ποιότητα ζωής και κοινωνική συνοχή. Εμείς τι κάνουμε, κάνουμε ε, συγκριτική έρευνα. Κάνουμε συγκριτική, ε, σύγκριση μεταξύ των πληροφοριών, ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε πώς αποδίδει κάθε χώρα και κατά πάσα πιθανότητα τα τρία προγράμματα, οι τρεις βασικές δραστηριότητες ε, ε, που ε, μας έχουν κάνει πιο γνωστούς είναι οι ευρωπαϊκές έρευνες που γίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και στην Νορβηγία και στις υποψήφιες χώρες μέχρι τώρα. Η ε, Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας που παρακολουθούμε την ε, ε, πρόοδο στη θέση, στις θέσεις εργασίας, η έρευνα για την ποιότητα ζωής όπου μιλάμε με πολίτες και στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Εταιριών όπου μιλούμε με διευθυντές επιχειρήσεων και έχουμε και ένα δέκτυο ανταποκριτών που μας επιτρέπει να έχουμε και δύο παρατηρητήρια στα οποία παρέχουμε ε, επικαιροποιημένες πληροφορίες συνεχώς, το παρατηρητήριο για την εργασιακή ζωή και ε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τις Αλλαγές, όπου εξετάζουμε τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, επικεντρωνόμενοι κυρίως στην αναδιάρθρωση. Παρακολουθούμε την απόδοσή μας με βασικούς δείκτες, να σας δώσω κάποιους επιγραμματικά και κάποια στοιχεία, γιατί βλέπω ότι η πρόεδρος θέλει να ολοκληρώσω, οπότε θα ολοκληρώσω. Ε, this year up to October in, 200... Ε, Μέχρι τον Οκτώβριο φέτος έχουμε αναφερθεί σε 230 έγγραφα πολιτικής, 55 από τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά και μας έχουν ζητήσει να παράσχουμε πάνω από 119 συνεισφορές σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις και φυσικά εφαρμόζουμε και τα προγράμματά μας για υψηλό επίπεδο ε, χρήσης ε, του προπολογισμού, να υπάρχει η κατάλληλη χρήση του προσωπικού μας ε, και φυσικά όλα αυτά είναι με βάση τους ελέγχους και την παρακολούθηση που γίνεται. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα του πώς χρησιμοποίησατε εσείς ε, το έργο μας ε, ως προς την νεολαία, ε, χρησιμοποίησατε τα όσα έχουμε διαπιστώσει εμείς στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και επίσης για την εγγύηση για την νεολαία. Για την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της οικονομικής διακυβέρνησης τα χρησιμοποίησατε στην έκθεση για τις πτυχές της απασχόλησης σε σχέση με την Τρόικα και τις χώρες στις οποίες υπάρχει μνημόνιο και επίσης το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε σχέση με την ε, ετήσια έκθεση ανάπτυξης και ε, όσον αφορά την αναδιάρθρωση χρησιμοποιήστε το έργο μας για παράδειγμα στην έκθεση για την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και επίσης την πρωτοβουλία στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους ε, όταν υπάρχει αναδιάρθρωση της ε, διοίκησης στην Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όσους χαράσουν πολιτική. Βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας από τους βασικούς ε, ε, θεσμούς που υποστηρίζουμε. Ε, μπορούμε φυσικά να σας παράσχουμε ομιλητές και εμπειρογνώμονες, έγγραφα σε περίπτωση που χρειαστεί και υπάρχει και ένα γραφείο στις Βρυξέλλες το οποίο είναι σε συνεχή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι οι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα και με τα χαρά θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε εδώ στο έργο σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι η Κρίστα Σέρλατζεκ η οποία είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, OSHA. Τα ψηφίσαμε στην Επιτροπή αυτή σήμερα. Μα ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα το θέμα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και ιδιαίτερος εδώ στο νέο κοινοβούλιο για να εξηγήσω το τι ακριβώς κάνει ο οργανισμός μας, ο ΩΣΑ, και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας για το μέλλον. Ιδρυθήκαμε το 1996 στο Μπιλμπάο μετά από απόφαση του Συμβουλίου. Είμαστε από τους μη τυπικούς οργανισμούς. Συνεργαζόμαστε με ένα διοικητικό συμβούλιο τριών πλευρών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Πολύ σημαντική για μας. Είμαστε μικροί, μικρός οργανισμός και φυσικά εξαρτόμαστε από την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτή είναι η δομή της όσα ε, από τρεις, ε, τρία μέρη αποτελείται το Διοικητικό μας Συμβούλιο και επιπλέον υπάρχει και ένα δίκτυο εστιακών σημείων σε κάθε κράτος μέλος. Επίσημοι εκπρόσωποι είναι αυτοί του οργανισμού μας ε, σε κάθε κράτος μέλος και διορίζονται από την εκάστοτε εθνική κυβέρνηση. Είμαστε υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνοι μάλλον, για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις εθνικές διαδικασίες. Για να σκεφτούμε όμως γιατί είναι τόσο σημαντική η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα του. Ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια και υγεία στην εργασία αλληλοσυνδέονται. Οι χώρες που έχουν μεγαλύτερα περιστατικά και ατυχήματα στη δουλειά είναι λιγότερο ανταγωνιστικότητες, ανταγωνιστικές. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχουν πολλά ατυχήματα, δεν γίνεται η βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει φυσικά να είναι στη δουλειά του και όχι στο νοσοκομείο ή στο σπίτι και να αναρώνει από κάποια ασθένεια ή από κάποιο ατύχημα. Στην Ευρώπη έχουμε 4.500 ε, μοιραία ατυχήματα και 2,8 εκατομμύρια άτομα χρειάζεται να παίρνουν ε, άδεια πάνω από τρεις ημέρες για να νερώσουν. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια μέρες εργασίες. Είναι λοιπόν σημαντικές, ε, σημαντικά τα αριθμητικά στοιχεία. Και πρέπει τα μέσα για τη βελτίωση της κατάστασης να είναι διαθέσιμα σε όλους. Εστιαζόμαστε κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλεται σταθερά το μήνυμα αυτό, ότι η ασφάλεια και η υγεία είναι καλή και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό για μας σε ό,τι αφορά και την υιοθέτηση του νέου στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και αν δεν κάνω λάθος συζητήσατε σήμερα το πρωί. Φυσικά έχουμε και εμείς τις δικές μας προτεραιότητες, τις δικές μας εσωτερικές στρατηγικές. Και αυτό πάντα εγκρίνεται από το τριμερές διοικητικό μας συμβούλιο. Να σας παρουσιάσω ποιες είναι οι προτεραιότητες μας αυτές εν συντομία. Καταρχάς, πρώτος τομέας. Η πρόληψη και η πρόβλεψη αριθμητικών στοιχείων και τάσεων. Αυτό μέσω μελετών βάσει τεκμηρίων, ενημερωτικών μελετών για τους ε, ηθήνοντες, τους πολιτικούς όπως εσείς, αλλά και για, αλλά για άλλες ομάδες όπως οι επιστήμονες και οι εμπρεγνώμονες. Οι μελέτες μας είναι οι μοναδικές που αφιερώνονται ειδικά στην ασφάλεια και στην υγεία σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Έχει γίνει μία μελέτη, τώρα έχει ξεκινήσει και μία δεύτερη και ξεκινάμε και μεγάλες μελέτες για το τι συμβαίνει μέσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και κάνουμε καινοτομική εργασία προκειμένου να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για το μέλλον. Επίσης, ποσοτικοποιούμε όλο και πιο πολύ το κόστος της ασφάλειας και της υγείας στην απασχόληση. Όλοι φυσικά γνωρίζουμε ποια είναι το ηθικό χρέος, η ηθική επιταγή για την διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρήσιμο είναι να χρησιμόμαστε και ποιο είναι και το οικονομικό κόστος. Και αυξάνονται οι επαγγελματικές ασθένειες, τις οποίες και θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα προκειμένου να υπάρχει και καλύτερη πρόληψη. Τρίτη προτεραιότητα. Εργαλεία για διαχείριση OSH. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζουμε τι χρειάζονται στη τελική ανάλυση οι επιχειρήσεις. Βοήθεια για την καθημερινή διαχείριση της ασφάλειας και της ε, υγείας. Στο Bilbao λοιπόν έχουμε πρακτικά παραδείγματα. Έχουμε καινοτόμεα εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία έχουμε και επωνομάσει όειρα. Τα εργαλεία αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των κρατών μελών και για τις ανάγκες του κάθε τομέα, ξεχωριστά. Επόμενη προτεραιότητα είναι η ευαισθητοποίηση. Και αυτό γίνεται σε πάρα πολλές πτυχές της εργασίας μας. Να αναφέρω μία εκστρατεία. Μόνο αυτή, γιατί έχω και χρονικό περιορισμό στην ομιλία μου. Είμαστε οργανισμός επικοινωνίας και αυτό αποτελεί τμήμα των βασικών μας εργασιών. Η εκστρατεία λοιπόν Healthy Workplaces να έχετε υπόψη σας ότι είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία που αφιερώνεται σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. είναι αποκεντρωμένη αυτή η εκστρατεία και την διαχειρίζονται τα σημεία τα εθνικά. Λάβατε κάποιες σχετικές πληροφορίες ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης υπάρχει και η εκστρατεία αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχουν ε, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείε, εθνικοί φορείς, αλλά και ΜΚΟ. Τελευταία πρωτοβουλία τελευταία μάλλον προτεραιότητα είναι η δικτύωση της ε, γνώσης. Ξεκινήσαμε το πρώτο ως wiki το καλοκαίρι για να υπάρξει καλύτερη δικτύωση σε όλη την Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη και να συμμετάσχουν οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο στη διαμόρφωση τέτοιων εργαλείων σε ό,τι αφορά τη δικτύωσή μας Προσπαθούμε να εμπλέξουμε όσους πιο πολλούς φορείς γίνεται προκειμένου να διαβιβάσουμε το μήνυμά μας. Κυρίες και κύριοι, τώρα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα έργο το οποίο και εκτελούμε κατά εντολή σας. Αναθέσατε κάποια κονδύλια για μία μελέτη για τις δημογραφικές ε, αλλαγές και προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μας προσέλαβε να κάνουμε την εργασία αυτή για σας. Θα σας παρουσιάσουμε τα σχετικά πορίσματα με την πάροδο του χρόνου, τα επόμενα χρόνια. Είναι σαφές ότι αν θέλουμε να φτάσουμε και να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης του 2020 σε ό,τι αφορά την ενεργό απασχόληση μεταξύ 20 και 64 ετών, πρέπει τώρα να λάβουμε δράση. Για να μην φεύγει ο κόσμος πιο νωρίς από την αγορά εργασίας, πριν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Και επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι οι πρεσβύτεροι, αν θέλετε, του μέλλοντος. Και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη εργασία για την πρόληψη. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά αυτή την ομάδα. Επίσης, άλλος, άλλη ομάδα στόχος αποτελούν οι μετανάστες. Η επόμενη εκστρατεία μας θα ξεκινήσει το 2016 και θα αναζητήσει τρόπους βιώσιμη διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού και παραμονής ε, των εργαζομένων στην αγορά εργασίας μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης. Εμείς από τον Μπιλμπάο θα χαρούμε να ερχόμαστε τακτικά στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώνουμε για το τι κάνουμε και πώς προχωρούν οι εργασίες μας του χρόνου ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τα εργαλεία αυτά που χρειάζονται και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τις εργασίες μας σε ό,τι αφορά τη μελέτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προγραμματίζουμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την διοργάνωση ενός συνεδρίου για να σας ε, παρουσιάσουμε ενδεχόμενε συστάσεις που θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες ε, στη δουλειά σας ως ε, πολιτικοί και νομοθέτες. Να σας διαβεβαιώσω κλείνοντας ότι είμαστε ένθερμοι σε ό,τι αφορά την συνεισφορά που μπορεί να έχει η δουλειά μας για την, για το μέλλον της Ευρώπης. Ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη μας και θα συνεχίσουμε την εργασία μας για να προωθήσουμε την ασφάλεια και την εργασία στους ε, χώρους απασχόλησης της Ευρώπης. Τονίζοντας το ότι αυτή η διάσταση της υγείας και της απασχόλησης είναι ιδιαίτερο σημαντική σε καιρούς κρίσης. Και γι' αυτό χρειάζονται λοιπόν ε, επενδύσεις αλλά και αξιόπιστα δεδομένα. Η όσα λοιπόν ο οργανισμός μας έχει θέσει ως βασικό στόχο της να μπορούμε όλοι να γυρίσουμε με ασφάλεια, ασφαλής σώη και χωρίς προβλήματα στη δουλειά μας κάθε μέρα μετά τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Τελευταίος ο πριν πριν ε, σας δώσω το λόγο, σε εσάς τα μέλη της Επιτροπής, είναι ο Μάντλεν Σέρμπαν, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ETF. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση που είναι μια ευκαιρία αλλά και τιμή και προνόμιο για μας να μοιραστούμε μαζί σας τι κάνουμε. Αφού οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην μοναδικότητα των οργανισμών που αντιπροσωπεύουμε θα πρέπει να σας πω ότι και εμείς είμαστε ιδιαίτεροι ε, όσον αφορά την ε, λειτουργία μας και θέλω να τονίσω στο τι είναι, ε, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης που έχει την έδρα του στο Τωρίνο το ETF, το 2014 είναι ιστορική χρονιά, όχι μόνο επειδή εορτάζεται ε, τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι καλό να θυμάται κανείς, αλλά και επειδή το 2014, μάλιστα αυτές τις μέρες, γίνεται συζήτηση και εορτασμοί όσον αφορά την ε, πτώση του τείχους του Βερολίνου. Πρόκειται για μια φάση όπου η πολιτική στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία και τη Γαλλία, πρόεδρος ε, Μιτεράν και Κολ, αποφάσισαν ότι ήταν καλό να δημιουργηθεί ένας οργανισμός για να υποστηριχθούν οι χώρες ε, στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις στην Ήπειρο, όπου ε, ε, έπρεπε να βρίσκονται ε, ιστορικά ε, εδώ και χρόνια, αλλά μόνο μετά την πτώση του Βερολίνου μπόρεσαν πραγματικά να ενωθούν με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τότε λοιπόν γεννήθηκε αυτό το ο οργανισμός, άρχισε να λειτουργεί το 1994 και γι' αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια με τον αδερφό οργανισμό Σεντεφόπ, γιατί ορισμένοι ε, αναφέρονται στο Σεντεφόπ που δουλεύει στο, για την Ευρώπη, ενώ το ETF που ε, δουλεύει εκτός Ευρώπης. Ποια είναι η διαφορά, θέλω να σας εξηγήσω. Το ETF δεν δημιουργήθηκε ως ένα τμήμα του ΣΕΝΤΕΦΟΠ που υπήρχε ήδη, αλλά η πολιτική τότε αναφέρθηκε εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο είπαν απλά ότι όχι. Δεν θέλουμε ένα πολιτικό μέσο που θα ασχολείται με τις χώρες εταίρους. Εμείς θέλουμε να οικοδομήσουν το μέλλον τους στις χώρες τους και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και ένα στους οργανισμούς αφιερωμένους σε αυτές τις χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά, αυτή λοιπόν είναι η ιστορική αναδρομή. Γιατί είμαστε τώρα διαφορετικοί, γιατί είναι ο διαφορετικό μόνος από τους τέσσερις οργανισμούς που δεν έχει τριμερή τριμερές διοικητικό συμβούλιο. Γιατί, γιατί οτιδήποτε κάνει εμπνέεται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αν διεξάγονται από αυτές τους οργανισμούς και άλλα, άλλα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμπνεώμεθα από τόσα συμβαίνουν στην Ευρώπη για να προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στις χώρες όπου λειτουργούμε, όχι για να επιβάλλουμε, γιατί η Ευρώπη ποτέ δεν επιβάλλει, αλλά για να τους ενημερώσουμε για το τι λειτουργεί στην Ένωση και ενδεχομένως να χρησιμεύσουμε ως έμπνευση για αυτούς ώστε να βρουν λύσεις πολιτικές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξη του του ανθρώπινου δυναμικού τους. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε σε τριμερέ συμβούλιο, ε, το θέμα είναι ποιοι αποτελούν το συμβούλιο. Πριν από 1,5 χρόνο ίσως να θυμάστε την αναθεώρηση της, της ε, του ιδρυτικού κανονισμού του ETF που εξέπνευσε το 2008. Έγιναν πολλέ συζητήσει λοιπόν και μία από αυτέ αφορούσε το ποιο θα πρέπει να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και το συμπέρασμα ήταν ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι παρόντα. Αλλά επιπλέον θέλαμε, και το Κοινοβούλιο το είπε αυτό, θέλαμε να έχουμε τρει ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε που δεν θα ψηφίζουν αλλά που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ETF πλέον από ε, των ε, τριών ε, παρατηρητών που αντιπροσωπεύουν τις χώρε εταίρου. Και είναι εδώ παρόσα και η νέα παρατηρητρία ε, από αυτούς που συμμετέχουν στο Δίκαιο Συμβούλιο. Καταρχήν λοιπόν, εφόσον είμαστε μέσα στο ε, κτίριο της μίας εκ των δύο δημοσιονομικών αρχής κάνουμε ό,τι θέλει να κάνει η Ευρώπη γενικώ. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε καταρχήν είναι να σχεδιάσουμε κοινό μέλλον σε αυτόν τον ε, πολύπλευρο κόσμο. Ε, το 2015, 90% της οικονομικής ανάπτυξης δεν προέρχεται από την Ευρώπη. Σε αυτό τον πολύπλοκο κόσμο που μόνο το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται στην Ευρώπη και γυράσκει κιόλα. Αυτό επίση που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι το 50% των δαπανών για τις κοινωνικές δαπάνες γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για το τι αναζητάει η Ευρώπη. Και όταν συζητάμε για το ότι η Ευρώπη συμβάλλει στην στην πολιτισμένη παγκοσμιοποίηση, αυτό βασίζεται στις αρχές που έχει η Ευρώπη, στις αξίες της για τη, υπέρ του ανταγωνισμού και της ε, συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω με λίγα λόγια τι ακριβώς κάνουμε ως ETF. Η πρόσβαση στις πληροφορίες υπάρχει, αλλά η παρακολούθηση της μετατροπής των πολιτικών είναι κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε είναι όπως το σχολείο, όπου τα παιδιά έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, υπάρχει το ίντερνετ, χρειάζονται ακόμα τους δασκάλους, ε, προφανώς ναι, γιατί χωρίς δασκάλους δεν μπορούν να δουλέψουν η δύναμη των εξωτερικών σχέσεων είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Σε όλες τις χώρες όπου λειτουργούμε θεωρείται προτεραιότητα το ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά πού ε, εμείς εργαζόμαστε. Καταρχήν στις υποψήφιες χώρες, στην περιοχή της διεύρυνσης, Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία, επίσης στη γειτονία που είναι ο Νότος, δηλαδή οπότε μιλάμε για τη Συρία, τη Λιβύη, την Τινησία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, είναι οι χώρες μας. Ε, δουλεύουμε στο Ανατολικό, ξέχασα να πω την, την και το Ισραήλ. Ε, επίσης δουλεύουμε στα ανατολικά τμήματα της Υπήρου μας όταν αναφερόμαστε στην Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, τη Λευκορωσία και αυτές είναι οι δικές μας χώρες. Ε, συνεργαζόμαστε με την Κεντρική Ασία και η Ρωσική Ομοσπονδία είναι χώρα εταίρος. Τι κάνουμε τώρα εκεί εμείς, ασκούμε πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου, μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες για τους πολίτες αυτών των χωρών να έχουν το μέλλον τους τους στις χώρες τους. Αυτό είναι ο ρόλος που μας ανετέθη από εσάς, από το Συμβούλιο και δουλεύουμε υπό τον άμεσο συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επειδή αναφέρθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να πω ότι η πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου είναι η Κομισιόν και αντιπροσωπεύεται από την DG ε, αλλά από την πρώτη πρώτου από την DG Απασχόλησης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, όπως είπα, είναι να δώσουμε μια ευκαιρία στους ε, ανθρώπους αυτών των χωρών να μείνουν στις χώρες τους και να αναζητήσουν το μέλλον τους στις ίδιες τις χώρες τους. Ε, προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες των πολιτών να βρουν δουλειά στις χώρες τους. Παραδείγματα, γιατί διαφορετικά είναι εύκολο να λέει κανείς θεωρίες για το τι κάνει. Θα ήθελα με την αδειά ε, σας, εκτός από το φυλάδιο που μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουμε. Ας πούμε όταν μιλάμε για δημόσια πολιτική είναι σημαντικό να έχουμε κοινή, ε, κοινό όραμα ε, στις χώρες. Μία σχετική διάσκεψη έγινε στην Αλβανία στις 6 Οκτωβρίου. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλες αυτές οι υποψήφιες χώρες είναι ότι οποτεδήποτε επενδύουμε κάτι σε αυτές τις χώρες, τους ζητούμε να δημιουργήσουν ένα έγγραφο στρατηγική. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά έχουμε πάρα πολλά χαρτιά, αλλά πολύ λίγη ε, εφαρμογή. Γιατί, γιατί όλοι, ε, μάλλον ο καθένα ακολουθεί τη δική του στρατηγική και δεν επενδύει απαραίτητο ότι θα πρέπει να γίνει εκεί. Και γι' αυτό στην Αλβανία, όπω και σε όλε τι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκάνιων, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τι απόψει των διαφόρων Υπουργείων και άλλων θεσμών σε ένα όραμα. Και αυτό, για παράδειγμα, βοήθησε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε στις 6 Οκτωβρίου, να αναδιαρθρώσει ολόκληρο το πρόγραμμα δράσης της κυβέρνησης και τον προϋπολογισμό της χώρας, ώστε να επενδύσει τρεις φορές περισσότερο για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου και να χρησιμοποιήσει το σύστημα παρακολούθησης που φτιάχτηκε ε, με τη δική μας βοήθεια για αιτήσιες εκθέσεις ε, σχετικά από τα Υπουργεία. Και αν υπάρχει ζήτηση, συνεργαζόμαστε και με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να γίνει αυτό σε τομεακό επίπεδο αλλά και σε ε, περιφερειακό επίπεδο και αυτό κάνουμε για παράδειγμα στην Ουκρανία. Ε, δεν, δεν έχουμε πολλές ε, γνώσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε περιφερειακό επίπεδο. Και όταν μιλάμε για περιφέρεια στην Ουκρανία, είναι πολύ καυτά τα θέματα αυτά σήμερα και γι' αυτό αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με μια από τις περιφέρειες της Ουκρανίας ώστε να φτιάξουμε ένα σύστημα για να αντιστοιχίσουμε τις δεξιότητες με τη ζήτηση σε περιφερειακό επίπεδο. Και τώρα οι υπόλοιπε περιφέρειες στην Ουκρανία προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα γίνει αυτό και είμαστε παρόντες για να τους βοηθήσουμε να γενικεύσουν το σύστημα αυτό σε όλες τις περιφέρειες. Το θέμα είναι τι κάνουμε όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Προσπαθούμε να την δημιουργήσουμε μέσω των δικών μας παρεμβάσεων στην ανάπτυξη την επιχειρηματική και περωθώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σε συνεργασία με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Ε, πολύ λίγα παραδείγματα, αλλά αν οι πολίτες από αυτές τις χώρες ε, γίνουν δεκτοί να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη μέσω της νόμιμης μετανάστευσης, εξασφαλίζουμε να έχουν ε, σαφής, σαφή προσόντα και πτυχία και να δουλέψουμε υπέρ της κυκλικής μετανάστευσης, ώστε αν επιστρέψουν στις χώρες τους η εμπειρία που έχουν κερδίσει στη διάρκεια της μετανάστευσής σας να αναγνωρίζετε. Αυτό είναι τμήμα της ε, συνεργασίας ε, με τις χώρες εταίρους. Είμαι στη διαθέσή σας και ευχαρίστως θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank all of you. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα θα ήθελα να σας δώσω το λόγο, να δώσω το λόγο στους υπολείπους δηλαδή, μπορείτε κάλλιστα να το ζητήσετε, αλλά θα ξεκινήσω Να ζητήσω όμως από τους συντονιστές πρώτα να λάβουν το λόγο, ο κύριος Κάσα καταρχάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους. Είναι καλό να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας για το τι κάνετε στους οργανισμούς σας. Κυρία Πρόεδρε, έχω μια πρόεδρε μια πρόταση. Επειδή έχουμε πάρα πολλά νέα μέλη εδώ στην Επιτροπή μας, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε επισκέψεις ε, στους οργανισμούς για να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καταλήλως τους οργανισμούς ε, για το έργο μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου όταν θα συζητήσουμε τις επισκέψεις μας ε, στην Ευρώπη αργότερα στη διάρκεια τη θητείας μας για την επόμενη πενταετία. Εγώ θα περιοριστώ σε μία ερώτηση, διότι έχω και άλλη συνεδριάσει και δυστυχώς θα πρέπει να φύγω. Ε, χαίρομαι που υπάρχει ένας Μαλτέζος συνάδελφος και κάθεται εδώ από την άλλη πλευρά της αίθουσας και θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω την ερώτηση μου στον καθηγητή James Καλέχα και θα το κάνω και στα Μαλτέζικα αν μου επιτρέπετε. Κύριε Καλέγια, προηγουμένως αναφερθήκατε σε προγράμματα μαθητείας και πραγματικά με εξέπληξε η παρατήρησή σας, διότι προσφάτως διάβαζα σε μια Βρετανική εφημερίδα ότι το, στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνονται μεγάλες επενδύσεις από την κυβέρνηση για προγράμματα μαθητείας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω και θα ήθελα να ξέρω και δύο λόγια παραπάνω για τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από αυτές τις επενδύσεις. Τι αποτελέσματα είχαμε. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν η Ευρώπη ακολουθήσει σε αυτά τα βήματα γιατί θεωρώ ότι τέτοιες κινήσεις βοηθούν την αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να απαντήσω και στα μαλτέζικα. Θα μιλήσω μαλτέζικα λοιπόν. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ερώτησή σας, διότι και εμείς στον οργανισμό μας ε, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Στις αρχές του έτους έγινε μια μεγάλη διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν διάφορες χώρες. Χώρες οι οποίες ε, ε, έχουν ε, ισχυρά ανεπτυγμένη την πτυχή της μαθητείας και κάποιες άλλες οι οποίες χρειάζεται να το επεξεργαστούν περισσότερο το ζήτημα. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, οι κάτω αλλά και άλλες, στις οποίες υπάρχουν εδρεωμένα προγράμματα μαθητείας ε, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά ε, ανεργία, κυρίως της ανεργία των νέων. Και γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά σοβαρό στην Ευρώπη, διότι έχουμε πάνω από 25 ε, εκατομμύρια νέους που αναζητούν θέση εργασίας. Και φυσικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν οδηγούν πάντα τους νέους στην πιο άρτια προετοιμασία για την αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν το οποίο διδαχθήκαμε από τις χώρες αυτές, χώρες όπως η Γερμανία, οι κατοχώρες και η Αυστρία, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς, είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές ευκαιρίες για τους νέους και μπορούν ε, πλέον να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία μαθητείας. Προσφάτως ε, έμαθα από τη Σουηδία συγγνώμη, από την Ελβετία διορθώνει ο ότι υπάρχουν 99.000 νέες θέσεις μαθητείας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις ε, που δημιουργούνται πλέον ε, για μαθητεία και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ε, για τους νέους και υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας χάρη ε, στην επίσημη κατάρτιση στην οποία ε, λαμβάνουν, στην οποία δεν θα είχαν πρόσβαση χωρίς τα προγράμματα μαθητείας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστούν καλύτερα για αυτά τα προγράμματα μαθητείας και να ασχοληθούν περισσότερο με τη μαθητεία, όχι μόνο ε, σε βιοτεχνικά επαγγέλματα, αλλά και για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουμε όλοι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να προσελκύσουμε περισσότερους νέους. Πολλές χώρες έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το θέμα αυτό. Εμείς, για παράδειγμα, στη χώρα μας έχουμε ήδη αρχίσει να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και προσπαθήσαμε να ε, προωθήσουμε τις ιδέες αυτές και να υπάρχει μαθητέα ήδη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε, επομένως, όταν ε, κάποιοι σπουδαστές δεν μπορούν να σπουδάσουν σε ανώτατα ιδρύματα, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, θα μπορούν χάρη στην μαθητεία σε μια επιχείρηση να μπορούν να μάθουν κάτι περισσότερο και να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός τρόπος να προχωρήσουμε και όσον αφορά την κατάρτιση και όσον αφορά την παιδεία για τους νέους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ε, χρησιμοποιείται η διαδικασία της μαθητείας και από πανεπιστήμια. Ευχαριστώ, η Γιούτα Στάινμπεργκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους οργανισμούς για τη δουλειά τους τα τελευταία πέντε χρόνια. Γνώρισα ποιες είναι οι διαφορές ε, σε ό,τι αφορά και την προετοιμασία των ε, εκθέσεων από πλευράς της ομάδας μου. Γι' αυτό λοιπόν αυτό και μόνο με κάνει να σας πω ευχαριστώ γιατί η ενεργεία των νέων είναι κάτι το οποίο καταπολεμείται μέσα από διάφορους οργανισμούς και το θέμα της διαβίου κατάρτισης και του δημογραφικού θέματος σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη των εξελίξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή για μας στην Ευρώπη να προβλέψουμε πώς θα αλλάξουν οι απαιτήσει της οικονομίας, της βιομηχανική παραγωγής στο μέλλον, προκειμένου εγκαίρους να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να απαντήσουμε. ξέρω και γνωρίζω κάθε οργανισμό προσωπικά και αυτό έχει μεγάλα πλεονεκτήματα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό για όλους τους συναδέλφους και για τους καινούργιους και για τους παλιούς συναδέλφους. Για το ETF. Για τον Ευρωπαϊκό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική ε, Εκπαίδευση. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι πραγματικά ε, ο κατεξοχήν τρόπο εκδημοκρατισμού του κόσμου. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι όλοι πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Υπάρχει και η πτυχή του κόστους. Και κάποιοι πιστεύουν ότι αν απαλλασσόμεθα από το κόστος των ατυχημάτων και των ασθενειών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήταν πιο ανταγωνιστικές. Εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρη, αλλά πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εφαρμοστούν διάφορα πρότυπα προκειμένου να υπάρξει πιο πολύ ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Είναι ρητορικό το ερώτημα, το γνωρίζω, αλλά ενδεχομένως να έχετε διεξαγάγει σχετικές μελέτες και έρευνες. Σε ό,τι αφορά το ΣΟΝΤΕΦΟΠ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα θέματα της ανεργίας των νέων, τα προσόντων των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασία και όλα αυτά. Πού πιστεύετε ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα προσκόμματα, τα μεγαλύτερα εμπόδια, γιατί υπάρχει τόσο αργή εξέλιξη στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Εγώ από τη Γερμανία γνωρίζω πάρα πολύ καλά το διτό σύστημα κατάρτισης. Και ξέρω ότι έχουμε προβλήματα παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το διτό σύστημα. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ απαραίτητο να υπάρχει υπάρχουν οι βέλτιστες ε, συνθήκες για τους νέους στην αγορά εργασίας. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να επιταχυνθεί αυτή η κατάσταση, αυτή η διαδικασία, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά το Eurofund τώρα, Eurofound. Συνεργαστήκαμε κατά το παρελθόν μαζί πάρα πολύ καλά. Και θα ήθελα να είχαμε συνεργαστεί σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της διαδικασία για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, γιατί έχετε την τεχνογνωσία. Τι πρέπει να αλλάξουμε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα και θα είχα άλλα τόσο να σας κάνω αλλά ίσως θα χρειαστεί να τα κάνουμε κατηδίαν αυτά τα ερωτήματα, να τα συζητήσουμε, μια και δεν έχω χρόνο. Um, for... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι αυτά που ο Επίτροπος για την εκπαίδευση συζητάει τα τελευταία χρόνια είναι η σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Και αυτός ο διάλογος θεωρώ ότι επί της αρχής μπορεί να φαίνεται σαν ένας εύκολος στόχος. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς συνδέουμε αυτούς τους δύο κόσμους, γιατί δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα. την ταχύτητα της αγοράς εργασίας και την ταχύτητα της εκπαίδευσης, η αγορά εργασίας πάει με χίλια δεν σημαίνει το ίδιο στην αγορά εργασία. Ποια είναι τα προσκόμματα, μα ρωτήσατε, τα εμπόδια. Μπορούμε να βελτιώσουμε την επαγγελματική κατάρτιση μόνο να κατανοήσουμε καλύτερα την αγορά εργασία. Αλλά αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και να περιορίζεται μόνο σε όσου ε, βρίσκονται στην αγορά εργασία. Θα πρέπει όλα αυτά να προσχωρήσουν στα επαγγελματικά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάω για προγράμματα μαθητείας, ανοίγουμε ένα ολόκληρο κόσμο σε νέους που προτιμούν να μαθαίνουν στην πράξη, σε μια επιχείρηση που μπορούσε, θα μπορούσε να τους προσελκύσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική κατάρτιση. κάνει τεράστια δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο εφαρμόζει και εγκρίνει μάλλον μεγάλο τμήμα της νομοθεσίας που αν εφαρμοστεί θα βελτιωθεί πολύ, πολύ, κατά πολύ την κατάσταση. Για παράδειγμα, άτυπη και τυπική εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι πολλές γνώσεις στην οικονομία μας παραμένουν κρυμμένες, δεν αναγνωρίζονται επίσημα. Δεν ε, μεταφράζονται σε προσόντα τα οποία μπορεί να διαβάσει, να επιλέξει ο εργοδότης. Φυσικά η έρευνα, η, συγγνώμη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της ενεργείας. Χρειάζονται και επενδύσεις. Χρειάζονται μια νέα πνοή της οικονομίας, προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις όχι μόνο στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, αλλά σε νέες θέσεις απασχόλησης, σε νέα προσόντα, σε νέες οδούς για πιο πολλές θέσεις απασχόλησης στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος που προσωπεί το to give the floor to uh, uh, another agency first. Αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο σε άλλη... Ε, ένα άλλο οργανισμό. Να απαντήσω στα γερμανικά. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και φυσικά... Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της νομοθεσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει και δική μας η μελέτη, ότι η νομοθεσία για παράδειγμα, οι επιθεωρήσεις μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την δραστηριοποίηση στην τομέα της προστασίας ε, της εργασίας. Όχι να υπάρχουν δηλαδή δύο μέτρα και σταθμά στην νομοθεσία. Όλοι θα πρέπει στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε από το διαδίκτυο δωρεάν και αποτελεί τεράστια βοήθεια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τέτοια εργαλεία που υποστηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις. Όταν μας λένε ότι μόνο οι επενδύσεις βοηθούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι μελέτες καταδεικνύουν το αντίθετο. Ένα ευρώ που επενδύεται αποδίδει δύο ευρώ. Αλλά αυτή η αναλογία φτάνει μέχρι και ένας προς δέκα. Εμείς στον οργανισμό μας έχουμε ξεκινήσει ένα project εδώ και πολύ καιρό, όπου προσπαθούμε να συνενώσουμε μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στις μικρές επιχειρήσεις για να υπολογίσουμε αυτή την απόδοση της επένδυσης. Προσπαθούμε να συγκρίνουμε λοιπόν την ε, εκαστοτέ απόδοση και ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή μέθοδο που θα επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρές επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των επενδύσεών τους. Να μην υπάρχουν λοιπόν δύο τάξεις, αλλά να υπάρχουν βοήθεια και υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τέτοια εργαλεία προκειμένου να βλέπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι πραγματικά αποδίδουν οι επενδύσεις τους. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μενέντες Βαλδές για την ε, μη τηλεμένη εργασία. Αυτό το θέμα το συζητήσατε και το πρωί. Είναι περίπλοκο. Όπως σας είπα, υπάρχουν διάφορα μέτρα για διάφορες καταστάσεις για να ελαχιστοποιηθούν οι διάφορες περιστάσεις σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ε, δήλωσης νέων ε, υπαλλήλων σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι υπάρχουν ε, διαφορά σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, τα κίνητρα, αλλά και πιο θετικά μέτρα, όπως πιο απλές διαδικασίες δήλωσης κτλ. Και για θέματα κινήτρων σε όσους δεν είναι δηλωμένοι. Ε, και εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια, ένα σωστό συνδυασμό μέτρων και κινήτρων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αξιολόγηση της πολιτικής. Εκεί είναι χρήσιμη η έρευνα. Εκεί μπορούμε να βρούμε τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Now it's Mr. Krasnodebski representing ECR. Uh, thank you very much. I will speak. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα πολωνικά. Κύριος Κρασνοντεύσκη. Έχω μια, ένα, μια παρατήρηση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στη χώρα μου και όταν συγκρίνω τα όσα λένε με τα όσα λέτε εσείς, συμπεραίνω πως υπάρχει μεγάλο, μεγάλη διαφορά γιατί η πραγματικότητα είναι δραματική στη χώρα μου τουλάχιστον όπου η κατάσταση είναι πραγματικά άσχημη. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση μέχρι στιγμής. Μεγάλη ε, διαφορά λοιπόν με τις δραστηριότητες των ε, οργανισμών σας, οι, οποίες, ε, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με πολύ καλά και θετικά λόγια. Ακούμε διάφορα για μελέτες, διασκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια κτλ. Και μάλιστα κάποιοι από τους οργανισμούς λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο πρέπει να καταπολεμήσουμε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση που αγγίζει όχι μόνο τους νέους αλλά και τους ηλικιωμένους που πολλές φορές έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις ε, χώρες τους για να αναζητήσουν την τύχη τους. Αυτό δεν σας ε, κάνει, δεν σας δημιουργεί, ε, δεν σας στεναχωρεί, αφού δουλεύετε σε τέτοιου είδους ε, οργανισμούς και επίσης ε, κάνετε κάποιο είδους εσωτερικό έλεγχο στις δραστηριότητε σας. Προβληματίζεστε για όλη αυτή την κατάσταση. Διότι βεβαίως τα όσα κάνετε δεν μπορούν να αναιρέσουν την κρίση, να εξαλείψουν την πηγή της, αλλά θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση σε κάποιες χώρες οι οποίες ε, ταλανίζονται από την ενεργεία εδώ και κάποια χρόνια. Παραθέσατε το παράδειγμα της Γερμανίας και της Αυστρίας και την σχετική επιτυχία της Γερμανίας και της Αυστρίας που δεν απορρέουν από το εκπαιδευτικό του σύστημα, αλλά από την οικονομία του. Η οικονομία τους είναι ισχυρή γιατί οι οικονομίες άλλων χωρών είναι αδύναμοι. Ίσως λοιπόν οι οργανισμοί σας θα πρέπει να στοχεύσουν διαφορετικά. Σε καιρού κρίση θα έπρεπε να ενεργήσετε ίσως μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω ποιο θέλει να μιλήσει για αυτούς τους προβληματισμούς. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο επικρατεί αυτή η σύγχυση στην οχυρία και πώς να την αντιμετωπίζετε. Όχι, εγώ δεν μιλώ για ασθενοχωρία, αλλά να σας δώσω ίσως ένα παράδειγμα. Βεβαίως μπορείτε να φανταστείτε ότι η ασφάλεια και η υγεία ε, δέχονται πιέσεις όταν έχουμε οικονομική κρίση. Είναι ένας από τους τομείς όπου οι εταιρείε. Οι εταιρείε σκέφτονται να μειώσουν το, πάντα το, τα κονδυλιά που προβλέπουν. Αλλά σας δώσω ένα θετικό παράδειγμα, όπως είπα και προηγούμενα, οργανώνουμε διετής εκστατείες για συγκεκριμένα θέματα. Ας πούμε, παράγουμε ενημερωτικό υλικό για το επίπεδο της εταιρείας, για ερευνητές, για πρακτικούς στις 25 γλώσσες αλλά και ε, εύκολα μέσα για μικρές επιχειρήσεις και στο Διοικητικό μας Συμβούλιο έχουμε τους εκπροσώπους 28 κρατών μελών. Και η ανταπόκριση που έχουμε ιδιαίτερα από χώρες που υποφέρουν από την οικονομική κρίση είναι ότι εάν εμείς δεν διοργανώναμε αυτές τις διετήσεις εκστρατείε. δεν παρήχαμε ενημέρωση, συστήματα και βοήθεια σε εθνικό επίπεδο δεν θα είχαν πια τίποτα. Δεν είναι η Γερμανία, δεν είναι η Αυστρία, δεν είναι ούτε οι κατοχώρες που μας ρωτούν. Ίσως ούτε οι βόρειες χώρες, αλλά οι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες πραγματικά μπορούν να ωφεληθούν. αυτό που κάνουμε τις, για τις χώρες ε, που είναι σε καλύτερη κατάσταση είναι να δίνουν το παράδειγμα και να βοηθούν στην ε, πλαίσιο της όσα ας πούμε για παράδειγμα να πάνε στις γειτονικέ χώρες και να βοηθήσουν ε, στον κοινωνικό διάλογο. Γιατί σε ορισμένε από τις χώρες αυτές βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τον εύρυθμο κοινωνικό διάλογο. Ξέρουμε πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει, αλλά τουλάχιστον αυτό το παράδειγμα για αυτή το είδο της εκστατείας δείχνει ότι μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τις χώρες που είναι υποπίεση. Σας ευχαριστώ. Μόνο ένα συντονιστή βλέπω ακόμα που δεν έχει Υποβάλλει ερώτηση. Θέλετε να υποβάλλετε ερώτηση, Τζιν Λάμπερτ, για αυτέ του οργανισμούς. Αν δεν θέλετε, έχω άλλου να που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ναι, λυπάμαι. Είχα ε, να ασχοληθώ με ιστορίες για, ε, για την κατασκοπία στις διασκέψεις για το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, έχω μια ερώτηση για ανθρώπους οι οποίοι ε, πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή ε, είναι εν εξελίξη η διαδικασία για την αναθεώρηση της μπλε κάρτας της σχετικής οδηγίας και υπάρχει και ένας οργανισμός ο οποίος εργάζεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάνει και πολύ καλές εκθέσεις στο παρελθόν ε, για την προοπτική των ανθρώπων για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ας ως προορισμό αν θέλετε, ως τη μοίρα τους για το άτομα υψηλών προσόντων και θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα για την έκθεση αυτή και τις εμπειρίες τους. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ναι, όντως, εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαστε με την κινητικότητα της εργασίας. Είναι τμήμα ούτως ή άλλως των θεμάτων που μας απασχολούν και αυτό που διαπιστώνουμε από την ανάλυση που κάνουμε σε όλες τις χώρες είναι ότι καταρχάς υπάρχει μια κινητικότητα από βορρά προς νότο και από νότο προς το βορρά, αλλά υπάρχει και από το νότο προς το νότο. Τι εννοώ με αυτό. Ε, συνήθως οι άνθρωποι από το νότο πηγαίνουν ε, προς τη Βόρεια Μεσόγειο, αλλά υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα ε, μεταξύ των χωρών. Πολλές χώρες, ε, πολλές από τους ανθρώπους της Νότιας Ευρώπης πηγαίνουν στις χώρες του κόλπου. Ε, τι γίνεται. Γίνεται και μεταφορά αντίστροφα. Δηλαδή από τις χώρες του κόλπου έρχονται εδώ. Το ίδιο ισχύει και από την ανατολική πλευρά του, ε, της ε, Ευρώπης. Οι πιο μορφωμένοι πηγαίνουν ε, προς την Ανατολή, δηλαδή ακόμα και στη Ρωσία, λόγω της γνώσης της γλώσσας. Το θέμα της γλώσσας είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Και το θέμα είναι ότι ο προορισμός των πιο καλά εκπαιδευμένων ανθρώπων δεν είναι απαραίτητο η Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά τώρα εδώ σχολιάζω το φαινόμενο. Από την άλλη, ε, το έργο μας ε, επιμένει στην κυκλική μετανάστευση, δηλαδή την ανάγκη των ανθρώπων να μετακινούνται. Δεν είναι κάτι βέβαια το οποίο θα πρέπει να σχολιάσω εγώ εδώ στην Επιτροπή σας, αλλά η μετανάστευση είναι και προσωπική απόφαση. Πολλές φορές οι άνθρωποι ε, μετακομίζουν σε μια άλλη χώρα για εργασιακούς λόγους. Η εργασιακή λοιπόν κινητικότητα ε, σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν ε, μακριά από τη χώρα τους ε, για πάρα πολύ καιρό. Θέλουν να επιστρέψουν, αλλά θέλουν να επιστρέψουν με την ανάλογη αναγνώριση και χωρίς να στιγματίζονται. Θέλουν να επιστρέψουν για ένα καλύτερο μέλλον. Και υπάρχουν δύο προβλήματα. Ε, συνεργαζόμασταν σε κάποιες από τις χώρες με ε, διεθνείς οργανισμούς μετανάστευσης που ε, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες που είχε δημιουργήσει ο οργανισμός μας ήδη ακόμα και σήμερα. Διότι εμείς είχαμε επικεντρωθεί στην προετοιμασία πρώτης αναχώρησης. Δηλαδή, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν και να μεταναστεύσουν νομίμως, καλό είναι να έχουν διαφάνεια στις δεξιότητες που έχουν επιτύχει και να είναι γνωστές και κατανοητές αυτές οι δεξιότητες στη χώρα προορισμού τους. Αν ε, αυτό είναι κατανοητό, τότε η χώρα προορισμού από εκεί και πέρα αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις δεξιότητες και τους ανθρώπους, διότι πρόκειται για ανθρώπων. Αλλά αν κάποιος θέλει να επιστρέψει, η χώρα καταγωγής τους έχει ένα μηχανισμό για να αναγνωρίσει την εμπειρία αυτών των ανθρώπων και να βεβαιωθεί ότι ε, υπάρχει και διασφάλιση ποιότητας. Και τι εννοώ με αυτό. Η αναγνώριση της εμπειρίας τους μπορεί να οδηγήσει στην απόφαση να τους δοθεί ένα επιπλέον δίπλωμα. Αλλά αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος διαφθοράς σε πολλές από τις χώρες αυτές, ακόμα και σε αυτές με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Και μπορεί να υπάρξει και μια ε, άνθηση, μια έκρηξη επιπλέον διπλωμάτων και όχι εμπειρίες που αποκόμισαν. Ε, αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε βέβαιοι σε αυτές τις χώρες ότι υπάρχει ένα σύστημα ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα μπορεί να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει με ποιοτικό, διάφανο τρόπο και να αναγνωρίσει δεξιότητες δεξιότητες και προσόντα είτε ε, στο εξωτερικό είτε στην ίδια χώρα ε, και να γίνεται με διαφάνεια για όποιον ενδιαφέρεται να ε, αναγνωριστούν τα προσόντα του. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε μαζί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας που πρόκειται για συμβατικές σχέσεις που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες από τις χώρες που έχουν υψηλό, μετανάστευση υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη. Και το θέμα είναι ότι στον αγώνα για τα ταλέντα κερδίζουν άλλοι και όχι η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σαρτιέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους, πολύ ενδιαφέρουσες. πολύ ενδιαφέρον και το έργο των διαφόρων οργανισμών και η έρευνά τους. Μία διαπίστωση, μία παρατήρηση και τρεις ερωτήσεις. Η διαπίστωση είναι ότι αναφερόμαστε σε προσόντα συνεχώς, αλλά λησμονούμε τον αριθμό των ε, προσόντων και των δεξιοτήτων στην κατάρτιση και ε, υπάρχουν και οι ανειδίκευτοι οι οποίοι ε, οδεύουν ολοταχώς προς την ανεργία και μάλιστα είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο κίνδυνος. Μόνο που οι άνθρωποι που είναι ανειδίκευτοι Ε, δεν αμφισβητεί, μέσω αυτών των ανθρώπων δεν αμφισβητείται μόνο η επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και η αρχική εκπαίδευση. Και αυτό σημαίνει ότι οι χώρες θα πρέπει να ανανεώσουν και να ξαναβάλουν στο σωστό δρόμο την αρχική έννοια της ε, εκπαίδευσης που έχουν, διότι πολύ συχνά αυτοί οι ανειδίκευτοι άνθρωποι έχουν ε, προβλήματα εξατομίκευσης του συστημάτων εκπαίδευσης, ε, διότι παντού στην Ευρώπη είναι ομαδοποιημένη η εκπαίδευση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε να δώσουμε νέα κίνητρα στα κράτη με Έλλη, να ε, βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανειδίκευτοι, δηλαδή να επικεντρωθούν στο σημείο στο οποίο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, παρατήρηση. Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με ε, τους οργανισμούς σας, συνεργάστηκα με πολλούς από εσά, κυρίως με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, για τις προβλέψεις απασχόλησης ε, νέες θέσεις απασχόλησης, ε, νέες δεξιότητες και πιστεύω ότι αφενός είναι σημαντικό να υπάρχουν προβλέψεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξισώσουμε την εκπαίδευση, την κατάρτιση με τις προβλέψεις, διότι ο χρόνος της κατάρτισης δεν είναι χρόνος εργασίας και αυτός που έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας και έχει μεγαλύτερο περιθώριο από ότι στην περίοδο της κατάρτισης. Τι θα προτείνατε στα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις προβλέψεις αυτές και να μπορούν να τις λάβουν υπόψη τους. Και τώρα, στις ερωτήσεις μου. Πού βρισκόμαστε σήμερα βάσει των αναλύσεών σας και των προβλέψεών σας ως προς την ε, ε, κατάρτιση με βάση τις δεξιότητες και όχι με βάση το περιεχόμενο. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά επικύρωση, την επικύρωση της εμπειρίας, της επαγγελματικής εμπειρίας, διότι τη συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και εξακολουθούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Ε, μιλάω ενώπιον ε, της, του πρώην Προέδρου της Επιτροπής μας, τον κύριο Άντερσον, και πραγματικά ε, ακόμα την ανανεώνουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η επαγγελματική κινητικότητα στην οποία αναφέρεστε περνάει από αυτή την επικύρωση, την πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας. Ιδάλλως βρισκόμαστε ακόμα στην ε, ακαδημαϊκή ε, εκπαίδευση και στην ε, άτυπη εκπαίδευση. Και επίση, ποιε είναι οι συνέπειε τη κρίση στη διαβίου μάθηση. Διότι βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε για μεγάλες επιχειρήσεις, ε, πιέζονται, αν θέλετε, λόγω της κρίσης, τότε η διαβίου μάθηση πάει περίπατο. Ο κύριος Μενέντης Βαλτές. Okay. Well, thank you very much for the question. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Νομίζω ότι πραγματικά ε, φτάσατε στον πυρήνα της υπόθεσης. Τέσσερα σημαντικά σημεία, λοιπόν μπορούμε να εντοπίσουμε για να έχουμε πιο πολλούς ανθρώπους που θα είναι έτοιμοι για να βγουν στην αγορά εργασίας. Το πρώτο θέμα λοιπόν που θέσατε είναι τι γίνεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τι γίνεται τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Φυσικά εδώ υπάρχει αρχή της επικουρικότητας. Κάθε κρατος μέλος είναι αυτόνομο, κάθε περιοχή είναι αυτόνομη και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Να μην ξεχνάμε όμως όπως πάντα αναφέρω, ότι όταν ε, ο κόσμος καταλήγει στην ε, επαγγελματική κατάρτιση, ουσιαστικά είναι αυτοί που δεν τα πήγαν καλά στην βασική εκπαίδευση, που δεν έχουν τα βασικά προσόντα. Όταν κάποιος δεν μπορεί να γράψει και να διαβάσει, δεν έχει καλή υποδομή σε ό,τι αφορά την πληροφορική, δεν μιλάει άλλες γλώσσες, έχει περάσει 11 χρόνια στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση αυτή. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε, θεωρώ. Και όχι να κοιτάμε πώς μπορεί η επαγγελματική κατάρταση να διορθώσει τα σπασμένα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για τη μείωση του αριθμού των μαθητών που φεύγουν πρόωρα από το σχολείο, αυτό θα είναι ένα φαινόμενο που θα συνεχιστεί. Θέλουν λοιπόν να βγουν στην αγορά της εργασίας, βγαίνουν για κανένα δύο χρόνια και δουλεύουν, αλλά μετά επανέρχονται στην επαγγελματική κατάρτιση χωρίς να έχουν όμως τα απαραίτητα προσόντα. Ύστερα, αν υπάρχει μια κατεπίγουσα ανάγκη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, δεν έχουμε χρόνο για τις προβλέψεις και δεν μπορούμε να Στριχθούμε αποκλειστικά σε αυτέ. Φυσικά οι προβλέψει είναι πάρα πολύ σημαντικέ ω δραστηριότητα και υπάρχει πάρα πολλή έρευνα η οποία κινείται προ την κατεύθυνση αυτή Τη πρόβλεψη των αναγκών τη αγορά εργασία. Αλλά έχουμε 9,4 νέου που ψάχνουν θέσει εργασία. Και έχουμε 2 εκατομμύρια θέσει εργασία που περιμένουν να πληρωθούν, να, να γεμίσουν. μπορούμε λοιπόν να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα αυτό είναι το θέμα. Και για να αναφερθώ σε αυτό που είπε πολύ ένα συνάδελφο πριν από λίγο. Είναι απογοητευτικό, αλλά αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός, να δούμε τι προβλήματα έχει ο Ευρωπαίος πολίτης και σε τοπικό επίπεδο, γιατί όπου υπάρχει ένα πρόβλημα υπάρχει και μια λύση. Η λύση λοιπόν αυτή σε μικρό, χαμηλό επίπεδο μπορεί να μην πρέπει ή μάλλον η λύση σε ένα πρόβλημα σε χαμηλό επίπεδο μπορεί να πρέπει να προέλθει από πιο υψηλό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις, αξιολογήσεις των προγραμμάτων μαθητείας. Έχουμε λοιπόν πιο λίγες χώρες φέτος, του χρόνου θα έχουμε τέσσερις χώρες, αυτό θα είναι μια βελτίωση. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση, πώς με ποια κριτήρια θα προσελκύσουμε πιο πολλούς για την απόκτηση τέτοιων προσόντων. Πολλοί αποθαρρύνονται και δεν ξεκινούν καν τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο. Αν οι διαδικασίες ε, αναγνώρισης δεν ισχύουν και δεν ε, εφαρμόζονται, αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο πρόβλημα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το 2016 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανανεώσουμε και θα ενημερώσουμε την αναγνώριση της ανεπίσημης και επίσημης ε, εκπαίδευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό σημείο, θετικό, θετική είδεση. Αυτό όμως ε, ωφελεί όλο το σύστημα. Πόσοι ωφελούνται η Γαλλία έχει ένα σαφές παράδειγμα για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και στην βάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι επιστημονική φαντασία αυτά που συζητάμε. Η εφαρμογή λοιπόν των ευρωπαϊκών εργαλείων, για να επανέλθω σε αυτά που έλεγα προηγουμένως, θεωρώ ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, το οποίο τα κράτη-μέλη δεν παίρνουν απαραίτητα εξίσου σοβαρά. Κάποιοι καθυστερούν σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν είναι το ίδιο με τα πανεπιστήμια. Κοιτώντα τι γίνεται στα πανεπιστήμια, πρέπει να πω ότι η όλη μεταρρύθμιση έγινε πολύ πιο γρήγορα. Τα πιο πολλά εργαλεία χρησιμοποιούνται στην ε, ανώτατη εκπαίδευση, όχι όμω στην επαγγελματική κατάρτιση. Μια τεράστια λοιπόν πρόκληση για εμά ω οργανισμό είναι το πώ. θα έχουμε πρόσβαση στα ιδρύματα επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν μιλάμε για μισό εκατομμύριο τέτοια ιδρύματα στην Ευρώπη. Τεράστια πρόκληση. Αυτή είναι η πρόκληση όμω που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, αν θέλουμε όντω να λύσουμε το θέμα του φαινομένου της εγκατάλειψη, τη πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου. Ευχαριστώ. Κύριε Καλέχα, Μαρίνο Ελπίντο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αγαπητή συνάδελφα, αγαπητή προσκεκλημένη. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και να ακούσω τη γνώμη σας για το τι γίνεται και το τι μπορεί να γίνει ώστε η ανθρώπινη εργασία να μην θεωρείται πλέον απλά και μόνο από οικονομική πτυχή, πλευρά, από την οικονομική πλευρά ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης, ως ε, παράγοντας κέρδους, αλλά να ε, εξετάζεται και ως ένας παράγοντας απελευθέρωσης του ίδιου του ανθρώπου, δηλαδή ένας παράγοντας επιβεβαίωσης της ελευθερίας του ατόμου και της ε, ηθαγένειας. Είμαστε στην Ευρώπη των πολιτών που θέλουμε να την οικοδομήσουμε και πιστεύω ότι η εργασία έχει κυρίως αξιολογηθεί από την οικονομική της πλευρά και θα ήθελα να ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί που εσείς ε, αντιπροσωπεύετε, ποια είναι η συμβολή που μπορούν να κάνουν ώστε να θεωρηθεί πλέον ως ένας παράγοντας ε, του ανθρώπινου όντως ως, ε, ως ε, ενός πολίτη, κυρίως στο επίπεδο της ισότητος. Ισότητος με γενικούς όρους και κυρίως ε, της ε, ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που οι γυναίκες συστηματικά αποκλείστηκαν από συγκεκριμένους χώρους εργασίας και από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης λόγω και μόνο ε, του ότι κάποια στιγμή θα γινούσαν. Υπήρξε μια τράπεζα που για χρόνια και χρόνια δεν δεχόταν υπαλλήλου γυναίκες επειδή θα έμεναν κάποια στιγμή έγκυε. Και σήμερα είμαι βέβαιος ότι οι γυναίκες πολλέ πολλές φορές πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην ε, δουλειά και την ε, μητρότητα. Να είναι δηλαδή γυναίκα πλήρω και να μπορεί να ε, ζήσει ως μητέρα, ως γυναίκα και να έχει και ε, πρόσβαση σε ένα επάγγελμα. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη, στη χώρα μου ε, και σε ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να ξέρω λοιπόν πώς μπορείτε εσείς να συμβάλλετε ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή νοοτροπίας στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στην Ευρώπη και κυρίως ε, εδώ μέσω των δικών σας οργανισμών. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους δύο τελευταίους που ζήτησαν να υποβάλουν ερωτήσεις. Και στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Είναι ο κύριος Λόπες και μετά ο κύριος Γιάνν Άντερσεν. Ωραία, τρεις ερωτήσεις, τρεις σύντομες όμως. Λόπες. Καταρχάς, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας και τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο και μία ερώτηση. Το σχόλιο για την παρέμβαση του κυρίου Καγιέχα για την τεχνική κατάρτιση και τις συνέπειες για την αγορά εργασίας. Και για να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα, στη χώρα μου, στην Ισπανία, η οποία ιστορικά έχει πολύ υψηλά ποσοστά ενεργείας, Σήμερα πλέον είναι σκανδαλώδη τα ποσοστά ανεργίας, αλλά ιστορικά είχε και υψηλά ποσοστά ε, φοιτητών πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ποσοστό σπουδαστών στο πανεπιστήμιο υψηλότερο από τη Γερμανία. Το πρόβλημά μας εδράζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει τεχνική κατάρτιση και αυτό έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και ε, το να υπάρχει μια γέφυρα και γι' αυτό είναι και η τεχνική εκπαίδευση σημαντική μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Ε, να σας πω επίσης ότι μπορεί να προκύψει η περίπτωση όπως συνέβη σε μας η αγορά εργασίας να είναι ε, ανασταλτικός παράγοντας για την τεχνική κατάρτιση εάν δεν έχουμε ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη στη χώρα μας ε, διαπιστώσαμε ότι εγκαταλείπουν περισσότεροι το σχολείο στις ακτές, στις παράκτιες περιοχές από ό,τι στην ενδοχώρα. Και ε, αυτό σημαίνει ότι δίνονταν ε, λανθασμένα μηνύματα και ήταν, θεωρούνταν ανασταλτικός παράγοντας η τεχνική κατάρτιση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Ε, ήταν πολύ σημαντική η παρουσίαση του Χουάν Μενέντεφ και έχει και κάποια σχέση με τις μελέτες του ε, για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασία που γίνονται σε μια σειρά από χώρε. Όπως γνωρίζετε ένα από τα μάντρα τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον στην ευρωπαϊκή δημόσια ε, συζήτηση είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα ήθελα να ξέρω τι συνέπειες θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε κάποιες αγορές εργασίας. Διότι αυτό το οποίο συνέβη είναι να αποδυναθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι συλλογικές ε, συμβάσεις, ε, να μειωθούν οι μισθοί προς τα κάτω πολύ, ε, σημαντικά και να υπάρξει και πολύ μεγάλο ποσοστό επισφαλών θέσεων εργασίας. Και αυτό φυσικά ε, θα ήθελα να ξέρω πώς θέλετε να τα συμπεριλάβετε στη συζήτηση για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, next question from, Επόμενη ερώτηση από την κυρία Σιντνάνσκα. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τους, ε, τους ε, καλεσμένους μας τι συγκεκριμένα μέτρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τι μπορούμε να κάνετε προκειμένου η επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση να αναγνωριστούν. Μιλάμε για μια τέτοια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά αυτές τις αγγίσεις. Μία δεύτερη ερώτηση. Πώς ε, πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα αυτά σύμφωνα με τις αναλύσεις σας. Είναι δύσκολο σήμερα να προβλεφθούν ποιες ικανότητες, ποια προσόντα θα χρησιμοποιηθούν και θα χρειάζονται σε 20 χρόνια. Όταν κοιτάμε τι γίνονταν πριν από 20 χρόνια, οι επιστήμονες δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει ποια ε, επαγγέλματα χρειάζονται σήμερα. Στις αναλύσεις σας λοιπόν, πώς επιλύεται το ζήτημα αυτό, το ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνουν τα παιδιά μας σε 20 χρόνια. Κύριος Άντερσον για την τελευταία ερώτηση. Δεν είναι πλέον βουλευτής, αλλά ήταν κάποτε, βουλευτή, ήταν κάποτε ε, πρόεδρος της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερως που βρίσκουμε και πάλι εδώ. Βλέπω κάποια γνώριμα πρόσωπα, αλλά και πολλά πρόσωπα που δεν αναγνωρίζω, πολλά καινούργια μέλη, πολλούς καινούργιους βουλευτές. Δεν θέλω να θέσω ερωτήσεις. Αυτό είναι δικό σας καθήκον ως βουλευτές. Να δώσω όμως κάποιες ε, σκέψεις ως συμβολή στη συζήτηση. Το Κοινοβούλιο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Είσαστε υπεύθυνοι για λήψη αποφάσεων και είσαστε και νομοθέτες. Για να ληφθούν λοιπόν αποφάσεις πρέπει να υπάρχει η σωστή γνώση για να μπορεί να είναι σωστή η απόφαση. Εδώ μιλάμε και έχουμε μαζί μα τέσσερι οργανισμού με πολλή εμπειρογνωμοσύνη. Μπορείτε να του χρησιμοποιήσετε του οργανισμού αυτού, πρωτού λάβετε τι αποφάσει σα και όλοι αυτοί. Γιατί έχω συνδεθεί με όλου αυτού και έχω σχέσει με έναν από του οργανισμού αυτού. Όλοι λοιπόν οι οργανισμοί έχουν σύνδεση άμεση με την αγορά εργασία και με, την θέση, με τις Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η πρόκληση για την Ευρώπη έχει να κάνει με την απασχόληση, με την ανεργία, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Και πιστεύω ότι ένα από τα κλειδιά, όχι το μοναδικό κλειδί, αλλά ένα από τα κλειδιά είναι η εκπαίδευση. Όλα τα είδη της εκπαίδευσης, στο σχολείο, το δημοτικό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη διαβίου εκπαίδευση. Από τη δική μου χώρα, τη Σουηδία το καθίσατε σαφές. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την πλειονότητα των κρατών. Να δούμε τι γίνεται με τους νέους σήμερα. Υπάρχει πολλή ανεργία. Αν συγκρίνουμε όμως τους νέους που έχουν την εκπαίδευση τη σωστή με όσους δεν έχουν εκπαίδευση και προσόντα, οι διαφορές είναι μεγάλες. Δεν είναι αυτόματο κλειδί η εκπαίδευση, αλλά είναι συνήθως καλύτερη θέση όσων έχουν προσόδα και έχουν εκπαίδευση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι νέοι που δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λοιπόν που συνδέεται και αυτή με την υγεία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, με τους όρους ε, που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Η Ευρώπη ποτέ δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί με κακά συστήματα εκπαίδευσης, με φτωχούς όρους εργασίας ε, στην αγορά εργασίας ή με κακούς μισθούς. Θα πρέπει να έχουμε το καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Θα πρέπει να έχουμε υψηλούς μισθούς και θα πρέπει να έχουμε καλή ασφάλεια και υγεία στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται. Γιατί οι εργαζόμενοι με την καλή εκπαίδευση θα έχουν και ψηλές απαιτήσει για το μισθό, για την υγεία και την ε, ασφάλεια. Άρα όλοι οι οργανισμοί αλλήλως συνδέονται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους οργανισμούς. Πριν λάβετε αποφάσεις, να έρθετε σε επαφή μαζί τους, όχι μόνο να, τις, να τους ακούτε, μια δύο στο χρόνο όταν έρχονται εδώ στην Επιτροπή, αλλά να έχετε επαφές μαζί τους. Για να λάβετε νέα στοιχεία, νέα γνώση για τα θέματα που πραγματεύονται. Γιατί είναι όλοι εμπειρογνώμονες, ξέρετε, ο καθένας στον τομέα του. Εγώ είμαι ένας από τους τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει το Κοινοβούλιο στο ETF στο Διοικητικό Συμβούλιο του ETF. Αξιοποιήστε με. Και εμένα και τους δύο συναντάλφους μου. Κρατήστε το email μου, τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Γιατί κάποιες φορές αναρωτιόμαστε τι γίνεται με τους οργανισμούς, τι θα γίνει με τους οργανισμούς αυτούς στο μέλλον. Είναι καλό να υπάρχει ανοιχτός διάλογος. Όταν μας διορίζετε, διορίζετε τρεις εμπειρογνώμονες, θα πρέπει να υπάρχει επαφή με σας. Στο Ευρωπαϊκό Έντρομα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχει και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, αλλά και τρεις εμπειρογνώμονες που έχετε ορίσει εσείς. Θα πρέπει να έχουμε δυνατότητες ανταλλαγής απόψεων. Τέλος για το ETF σε ό,τι αφορά τα θέματα μετανάστευσης. Έχουμε μετανάστευση και στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και από το εξωτερικό της Ένωσης προς την Ένωση. Και αυτό στο μέλλον θα οξυνθεί. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να κλείσουν τα σύνορά τους. Δεν ξέρουν τίποτα. Ο κόσμος είναι ανοιχτός. Και αυτό δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα. Υπάρχει, ναι, και μια πτυχή προβληματική. Υπάρχουν προκλήσεις αλλά και δυνατότητες που ανοίγει η μετανάστευση. Αυτό σε σχέση με αυτά που είπε η συνάδελφος, ρώτησε το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα προσόντα όσων έρχονται εκτός ε, από το εξωτερικό της Ένωσης. Έχουμε τη δημογραφική τάση, χρειαζόμαστε πιο πολλά άτομα και θα χρειαζόμαστε πιο πολλά άτομα στο μέλλον για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Χρειαζόμαστε λοιπόν άτομα, νέα ροή ατόμων από το εξωτερικό της Ένωσης, να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους για να υπάρχει ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης. Αλλά σας ζητώ επισταμένως να έχετε πιο πολύ επαφή μαζί μας. Μου άρεσαν πάρα πολύ ε, οι μήνες που πέρασαν εδώ πέρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ε, ο καλύτερος χρόνος της ζωής μου. Αλλά χαίρομαι επίσης που είμαι ένας ανεξάρτητος ε, εμπειρογνώμονας πλέον και θα ήθελα να σας βοηθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για Άντερσεν και τώρα θα σας δώσω τρία λεπτά στον καθένα. Από δεξιά προς αριστερά θα πάρετε το λόγο. Αν ε, ξέχασε κάποιος συνάδελφος κάτι, μην ξεχάσετε να το συμπληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ε, ο Πορτογάλος ε, Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη σημασία της εργασίας, του έργου και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Υπάρχει πολλή έρευνα που βασίζεται και στα ευρωπαϊκά αιτήματα, αλλά υπάρχουν και όλες αυτές οι ε, ρυθμίσεις τις οποίες βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή μπορεί να είναι προς όφελος της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας αλλά και των ίδιων των εργαζομένων. Και πολλά από αυτά δεν έχουν καμία σχέση ε, με ε, τα θέματα αυτά. Μας ενδιαφέρει η αυτονομία των εργαζομένων. Ε, προσπαθούμε να διευκολύνουμε ο, τους εργαζομένους ώστε να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους και δεν υπάρχει καμία σχέση με κόστος. Ε, ε, γίνεται πολλή δουλειά και σε αρκετούς οργανισμούς εργαζόμαστε ώστε να δώσουμε κάποια παραδείγματα για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και αυτές τις πτυχές. Επίσης, ε, είπαμε πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας των νέων ή και των γυναικών που αναφέρθηκαν. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Λόπεθ, θα σας απαντήσω στα ισπανικά. θίξατε διάφορα ζητήματα. Η σχέση της αγοράς εργασίας και της ε, κατάρτισης, να σας πω ότι υπάρχει ε, συσχέτιση άνω του 60%, 65% ε, μεταξύ των σπουδαστών που εργάζονται στη διάρκεια των σπουδιών τους ε, και ανθρώπων που έχουν ε, μια σταθερή σχεδόν σχέση εργασίας μετά από ένα χρόνο από την περάτωση των σπουδών τους. Και επίσης όσον αφορά των αλλαγών, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τις συλλογικές συμβάσεις, ε, να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μία καμπή και η πρόκληση είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο το στόχος και ακριβώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η ποιότητα της εργασίας είναι κατάλληλη, γιατί και αυτή είναι σημαντική, διότι οι συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε σήμερα θα μας οδηγήσουν σε βιώσιμες θέσει εργασία στο μέλλον και δεν θα, πρέπει, δεν θα θέλει να πρόωρα την αγορά εργασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε ε, τους στόχους ε, της απασχόλησης και του ποσοστού απασχόλησης και να αντιμετωπίσουμε και τις δημογραφικές προκλήσεις. Και μία τελευταία αναφορά στο σχόλιο του κυρίου Άντερσαν για το ε, παγκόσμιο ανταγωνισμό, που είμαστε ανταγωνιστικοί, ε, συνθήκες εργασίας, μισθή και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ερευνούμε επίσης. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνθήκων Εργασίας που κάνουμε αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 23 χώρες και θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες ε, ε, σε σχέση με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, την Κίνα, ήρθαμε σε επαφή με τις ΗΠΑ γιατί είναι πολύ καλό για την Ευρώπη να γνωρίζει βάσεως ανταγωνίζεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό σημαντικά στοιχεία ε, των εργασιακών σχέσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καγέχα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Δεν έχω κάποια άμεση λύση να σας πω. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία 10 χρόνια είναι να επισημάνει την αρχή της ίσης ε, ε, αξίας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της εμπειρίας που αποκομίζει κάποιος από επαγγελματική κατάδυση σε ένα τεχνικό επάγγελμα. Στις χώρες μου ή στην Ισπανία ή στη Μάλτα οι γονείς ε, πιέζουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. εάν γίνεις ανθρωπολόγος, γιατρός, δικηγόρος κλπ. θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στο σπίτι για να το γιορτάσουμε το πτυχίο σου, αλλά την άλλη μέρα το πρωί δεν θα έχεις δουλειά. Επομένως, οι αγορές εργασίας θα πρέπει να διεισδύσουν καλύτερα στην εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να κάνουμε κατά πάσα πιθανότητα, ώστε η αγορά εργασίας να προβάλλεται όσο το δυνατόν περισσότερο, το συντομότερο δυνατόν. Δεν αναφέρουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι κάποιοι αναφέραν ότι ακόμα και αυτή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται το πρώτο βήμα προς την αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μπορούν να ε, περάσουν στη, διαβίωση, στη διαβίου μάθηση στα 16, στα 18 τους με το σκεπτικό ότι πρέπει να αποκομίζουν δεξιότητες. Ό,τι δουλειά και αν κάνει κάποιος στο μέλλον, αν είναι σε οδηγό, ε, καθηγητής ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχεις ε, βασικές δεξιότητες που θα σου επιτρέπουν να χρησιμοποιείς τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία είναι η γλώσσα του σήμερα, πολλό δε μάλλον του αύριο, και αυτή η δυνατότητα είναι αυτή η οποία θα μας βοηθήσει να πιέσουμε το εργατικό δυναμικό μας στα επίπεδα ανταγωνιστικότητας στα οποία αναφέρετε κι εσείς. Βεβαίως και οι προβλέψεις μας λένε ότι τα επόμενα 10-20 χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε μεσαία τάξη δεξιότητα. Μεσαία τάξη δεξιότητα είναι δεξιότητε οι οποίε δεν απαραίτητο πτυχία. Και πώς μπορούμε να πείσουμε τους γονείς ότι τα παιδιά τους ε, σε 15-20 χρόνια δεν θα χρειάζονται ένα πτυχίο, αλλά με ένα δίπλωμα κατάρτισης θα μπορούν να εργαστούν. Και αυτή είναι η πρόκληση και αυτό είναι απογοητευτικό γιατί δεν μπορεί να τα πει κάποιος δημοσίως αυτά. Αλλά αν καταφέρουμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν στην ε, πιστοποίηση της άτυπης εκπαίδευσης. Είναι μια σύστοση του 2012. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτά που έχουμε, τις τομεακές δεξιότητες θα πρέπει οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι ε, και οι εκπρόσωποι τους να ε, συμπεριληφθούν και αυτοί στην ίδια εξίσωση και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, συγκεκριμένη εμπειρία και δεν έχουν κάτι να δείξουν ως αντάλλαγμα για την απασχολησιμότητά τους θα πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Θα σταματήσω εδώ γιατί τελείωσαν τα τρία μου λεπτά. Η κυρία Σέτετσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω διότι πολλά ακούστηκαν ήδη. Και να σας παραπέμψω και λίγο στο πρόγραμμα το οποίο εκτελούμε εξ ονόματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μεγαλύτερη ηλικία εργαζόμενοι και ασφάλεια και υγεία στον χώρο τη εργασία. Και θα ήθελα να σταθώ και στην απασχολησιμότητα, διότι εμεί θέλουμε να έχουμε ανθρώπου οι οποίοι θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά υγιεί στη θέση εργασία του. και επίση θα πρέπει να φροντίσουμε και του νέου ανθρώπου Και αναφέρθηκε και αυτό και οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν του κινδύνου, θα πρέπει να γνωρίζουν ε, θέματα που αφορούν τη δική του ασφάλεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Για παράδειγμα, μία από τις ανακοινώσεις μας και ένα μέσο πρόθεσης είναι μία εργαλειοθήκη για διδάσκοντες μέσω της οποίας τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τους κινδύνους και την ασφάλεια και να μπορούν να φροντίζουν να είναι υγιείς. Όσον αφορά τη διαβίου μάθηση, όπως σας είπα στο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε, έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε και με κάποιον εξωτερικό εργολάβο και η διαβίου μάθηση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ε, συλλέγουμε και πρακτικά παραδείγματα από όλα τα κρατημέλη και βλέπουμε ότι επιχειρήσεις οι οποίες είναι οικονομικά επιτυχής, ε, οι ευφυείς επιχειρήσεις ε, πολύ συχνά σε μεγάλες χώρες δεν σταματούν την εκπαίδευση ακόμα και στα 45. Συνεχίζουν μέχρι την συνταξιοδότηση και ένα παράδειγμα είναι η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, όπου μπορεί κανείς να βρει και προσφορά ε, στους εργαζομένους για να μείνουν μέχρι τα 70 τους και υπάρχει συνεχής επιμόρφωση η οποία φυσικά υποστηρίζει και την απασχολησιμότητα και την εργασία. Εμείς στην OSHA, ε, όταν επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια και στην υγεία, στην εργασία, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στους αναδυόμενους νέους κινδύνους, παραδείγματος χάρη, ε, ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, ε, αλλά επίσης και μειοσκελωτικές ασθένειες, οι, οποία είναι, οι οποίες είναι από τις ασθένειες που εμφανίζονται υψηλά στις ε, επαγγελματικές ασθένειες, και βρίσκονται και στην ε, ε, κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Είναι λοιπόν στοιχεία στα οποία θα πρέπει ε, να σταθούμε και θα πρέπει να εξετάσουμε και θέματα πρόληψης μυοσκελετικών ασθενειών. Τέλος, οι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εξετάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο σε εθνικό επίπεδο και σε τομεακό επίπεδο οι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν συνδρομή και στις καθημερινές τους εργασίες αλλά και στη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας και θα μπορέσουμε να σας δώσουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες αλλά να σας πούμε επίσης ε, που υπάρχουν λήψεις και περισσότερες απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα. Ε, 2015 και 2016 αυτά. Ευχαριστώ κυρία Σέρπαν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλά πράγματα συζητηθήκαν εδώ σημαντικά και θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής της προηγούμενης ειτίας γιατί συνέβαλαν πολύ στην ανάπτυξη των θεσμών στις χώρες εταίρους ε, και όπου δηλαδή λειτουργεί το ETF. Πραγματικά ελπίζω πως θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Όταν αναφερόμαστε στο τι κάνουν οι χώρες εταίροι, δηλαδή προσπαθούν να οικοδομήσουν τις δημοκρατικά πολιτεύματα, χρειάζεται να έχουν ε, κοινοβούλιο. Βέβαια, πώς θα το ονομάσουν ακριβώς είναι δικό τους θέμα, αλλά προς έκπληξή μας, και αυτό συνέβη στις αραβικές χώρες, πιστώσαμε ότι καμία από τις χώρες δεν έχει επιτροπή που να είναι αφιερωμένη στην απασχόληση. Θα ήταν καλό Εφόσον εσείς διαλέγετε τη συμμετοχή σας στις διάφορες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, να έχετε υπόψη ότι με τη βοήθεια που δίνουμε σε αυτές τις χώρες, σε αυτόν τον τομέα, ίσως να συμβάλλουμε και στο να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων θα είναι μέρος της ατζέντα τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και περάσατε κάποιες ώρες μαζί μας. Ε, κάνατε πολύ καλή εντύπωση. Ε, δεν νομίζω πως είμαι η μόνη που είμαι έτσι θετικά εντυπωσιασμένη μετά από τη συζήτησή μας. Θα είμαστε διαρκώς σε επαφή όπως ανέκαθεν και ίσως τώρα με τα νέα μέλη που έχουμε να έχουμε ακόμα πιο εντατικές επαφές. Και φυσικά προσπαθούμε να επισκεφθούμε όλους τους οργανισμούς που έχουμε, οπότε αργά ή γρήγορα θα έρθουμε να επισκεφτούμε και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συμβολή σας και σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Item 16, uh, the Russian embargo. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το 16, το ρωσικό εμπάργο, αν δεν κάνω λάθος. Στις 24 Σεπτεμβρίου οι συντονιστές αυτής της Επιτροπής αποφάσισαν ότι το θέμα του της επιρροής ε, στην οικονομία και την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ρωσικού Εμπάρκου θα ήταν ένα θέμα που θα συζητήσω στην Επιτροπή μας και αυτό θα κάνουμε τώρα. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Έκερτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Βεβαίως, ε, Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι λιγότερο ευχάριστο από το να δούμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις μελλοντικέ γενναίες. Μιλάμε για την απαγόρευση εισαγωγών από πλευράς Ρωσίας των ευρωπαϊκών προϊόντων και των τροφίμων. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό αν αν και σε ποιο βαθμό ο Ευρωπαϊκός, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί ο φόρτος ιδιαίτερα στη γεωργία και στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Να θυμίσω πως αυτό το εμπάργο που πλευρά Ρωσίας είχε μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά των ε, γεωργικών προϊόντων ε, γιατί ότι μεγάλο ποσοστό της αγροτικής παραγωγής αλλά και το 4,2 των αγροτοδιατροφικών προϊόντων επηρεάζονται. Οι εξαγωγές μας πολλές φορές ε, κατευθύνθηκαν προς την Ιαπωνία, την Κορέα και τις Φιλιππίνες, ωστόσο σε άλλους τομείς ε, ο αντίκτυπος ήταν πολύ σημαντικός. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για τα τρόφιμα και τα λαχανικά, όπου η Ρωσία αντιστοιχούσε περίπου στο 40% των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Να μιλήσω τώρα για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε το 2006 ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην απασχόληση. Επίτα επεκτάθηκε ώστε να καλυφθεί η οικονομική και δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και αυτό αντικατοπτρίζεται στον κανονισμό τόσο στο άρθρο 2 όσο και στο ε, ναι, κανονισμό. θα πρέπει επίση να διευκρινίσω ότι το EGF, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, δεν είναι ένα ταμείο που ε, καλύπτει τις απώλειες ε, εισοδημάτων, αλλά εκεί όπου έχουν γίνει σημαντικές ε, μεγάλες απολύσεις να μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους άνεργους. Δεν είναι δηλαδή ένα αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλεια εισοδήματος. Αν κανείς δει τα δύο κριτήρια, παγκοσμιοποίηση και κρίση, το κριτήριο για την κρίση δεν ισχύει βέβαια εδώ γιατί είναι οικονομική και, κοινο... οικονομική κρίση ε, που συνεχίζεται από το 2007-2008 ε, καλύπτεται από το EGF αλλά όχι το εμπάργκο το ρωσικό. Αυτό που θέλουμε περισσότερο να εξετάσουμε είναι κατά πόσο οι διατάξεις ε, στη στο, στο άρθρο 2α θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, γιατί εκεί γίνεται λόγος για τα κριτήρια παγκοσμιοποίησης, γίνεται λόγος για αλλαγές στο εμπορικό, εμπορικές συνήθειες και απώλεια τμήματο της αγοράς. Όταν εξετάσαμε μαζί με την νομική μας υπηρεσία στο θέμα περισσότερο, είδαμε ότι η πρόθεση αυτή τη διατύπωση αφορά την παγκοσμιοποίηση και ότι τα κριτήρια μεριδίου αγοράς, απώλεια μάλλον μεριδίου τη αγορά αφορούν και είναι δείκτε ώστε να αποδείξουν την επιρροή τη παγκοσμιοποίηση, ενώ η ρωσική, το ρωσικό εμπάργο δεν είναι συνέπεια παγκοσμιοποίηση από νομική άποψη, αλλά και από οικονομική άποψη, είναι το αντίθετο διότι πρόκειται για μια μονομερή απόφαση που πυροδοτήθηκε από μια άλλη μονομερή απόφαση για απαγόρευση των εισαγωγών από την Ένωση. Άρα λοιπόν δεν πληρείται το κριτήριο της παγκοσμιοποίησης και κατά συνέπεια το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να καλυφθούν οι επιπτώσεις αυτού του εμπάργου, ιδιαίτερα στον τομέα των αγροτοδιατροφικών που επιπλέον θα έπρεπε να αποδείξει μάλιστα απώλειες άνω των 500 εργαζομένων και όχι μόνο απώλεια εισοδήματος ή μεριδίου αγοράς. Αυτό θα είναι επιπλέον δηλαδή. Πάντως το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το EDF δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ, σε αυτή την περίπτωση και βέβαια η Κομισιόν λαμβάνει διάφορα ε, μέτρα στον τομέα της ε, γεωργικής πολιτικής σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης των διαφόρων αυτών ταμείων. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ανάλυσης που κάναμε και μετά από το αίτημα και τα ερωτήματα του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Άκουσα την ε, εξηγήση που μα έδωσε η Κομισιόν. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω ακόμη μια φορά την προσοχή σας στο γεγονό ότι οι βαλτικέ χώρες χτυπήθηκαν περισσότερο από το ρωσικό Ε, Εφόσον είναι λοιπόν ιστορική, ιστορικά ε, παράδοση, ε, η παραγωγή του τομέα αυτού να προορίζεται στη Ρωσία που είναι ο άμεσος μας γείτονας. Με τον και έχουμε και ιστορικούς δεσμούς. Οπότε η παραγωγή μας και η αγροτοδιατροφική βιομηχανία υπέφεραν πάρα πολύ. Οι απώλειες θέσεων εξακολουθούν να ε, γίνονται, να υπάρχουν ε, κυρίως στις γεωργικές περιοχές και για να δημιουργηθεί η εναλλακτική επασχόληση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έτσι ξεκινά ολόκληρη αυτή η αλυσίδα. Ο κόσμος κάνει τη δουλειά του, βρίσκεται κοινωνικά αποκλεισμένο. Ή μπορεί και να επιλέξει ακόμα χειρότερο σενάριο. Να φύγει τελείως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να θέλει και η Λουθανία να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να δούμε αν ε, γίνεται να χρησιμοποιηθεί το EGF για να βοηθήσουμε τους γεωργίους μας. Αλλά λάβαμε την απάντηση που ήταν σύντομη και πολύ τυπική. Λες και δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί. Ναι, κατάλαβα ποιες είναι οι διατάξεις, κατάλαβα ποιος είναι ο σκοπός του EGF και θυμάμαι και στην προηγούμενη θητεία το είχαμε συζητήσει για το αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο σε περιπτώσεις κρίσης κτλ. Καταλαβαίνω τις εξηγήσεις που μας δώσατε για το ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί αυτό το ταμείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ε, λύση. Γιατί τι άλλο είδος ε, τα κονδύλια και χρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το πρέπει να απαντήσουμε. Το ρωσικό εμπάργκο επί των προϊόντων των, της Ένωσης δεν είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, αλλά μιλάμε για πολιτικής φύσης μέτρα, συνέπεια ε, μιας πολιτικής κρίσης. Και αυτή είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο γείτονας ε, με την τελείως απρόβλεπτη συμπεριφορά είναι σημαντικό εταίρο. Θέλω να ζητήσω από την Κομισιό να το εξετάσει αυτό, όχι με την τυπική πλευρά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EGF, αλλά πρέπει να αναζητηθούν άλλοι πιθανοί ε, πόροι για να στηρίξουμε τους γεωργούς μας και μάλιστα πόροι που να μπορούν να κινητοποιηθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί ο κόσμο υποφέρει πολύ. Ζητώ την κατανόησή σα, διότι η κατάσταση είναι τραγική και θα πρέπει γρήγορα να βρούμε έναν τρόπο για να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να αναφέρω ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ήταν ε, μία από τις, από τις λίγες πολιτικές επιλογές που είχαμε μετά από την κατοχή της Κρυμαίας από τη Ρωσία και από την ε, ε, ε, υπόλοιπη συμπεριφορά της Ρωσίας. Δυστυχώς δεν ήταν λογική η ανταπόκριση της Ρωσίας στην Ουκρανία μέχρι στιγμής. Ωστόσο, διαπιστώνουμε μέτρα κατά κάποιων ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων. Και πάλι τα κυρώσεις αυτές δεν είναι η πιο επιθυμητή επιλογή στη σύγχρονη άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικονομική ανάπτυξη, μάλλον έχει περιορισμένες επιλογές σε τέτοιες καταστάσεις. Το οικονομικό μας συμφέρον δεν θα πρέπει να κυριαρχήσει σε αυτή την περίπτωση επί του ασφάλεια και των πολιτικών αρχών και αξιών μας. Δύο-τρία ερωτήματα στην Κομισιόν και μετά η Κομισιόν μπορεί να σχολιάσει την συνεχιζόμενη ε, εξέλιξη υποθέσεων κατά τη Ρωσία στον ΠΟΕ. Επίσης η Κομισιόν ετοιμάζει αξιολόγηση το, της του παγκόσμιου αντικτύπου της ύφεση στις ευρωπαϊκές χώρες και τι είδους οικονομικοί, ποιοι μάλλον οικονομικοί τομείς, σύμφωνα με τη γνώμη της Κομισιόν, ε, κινδυνεύουν περισσότερο μακροπρόθεσμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του εμπάργου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Στέβες Πιέτρο. Κύριε Κουτιέρης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συζητούμε τελικά ποιο πληρώνει την ύφη. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις για τους ε, ε, γεωργούς ε, στην Ευρώπη που πλήγησαν από το εμπάρκο της Ρωσίας. Και αποζημιώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες ακριβώς διότι οι Ευρωπαίοι γεωργιές δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τις συνέπειες της πολιτικής προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διεθνούς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι εγώ χαίρομαι για την παρέμβαση που ακούσαμε σήμερα από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην Επιτροπή Επασχόλησης, γιατί και εγώ ε, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να δώσει αποζημιώσεις στους γεωργούς. Ε, θυμάμαι ότι στη συζήτηση που κάναμε στην προηγούμενη θητεία πολλά μέλη της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας εδώ θέσαμε τις επιφυλάξεις μας ε, ένα ταμείο που είναι πολύ περιορισμένο και είναι ένα ε, ταμείο προσαρμογής ε, στην παγκοσμιοποίηση να χρησιμοποιείται και σε άλλους τομείς, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία που έχουν τρόπους χρηματοδότησης από την κοινή γεωργική πολιτική. Εδώ λοιπόν γίνεται μια συζήτηση ουσίας η οποία θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου. Είναι απαραίτητο οι γεωργοί να λάβουν αποζημιώσεις, ναι, ε, και μάλιστα πρέπει να γίνει τώρα, γιατί πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις, πολλές μικρές επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν είναι οικονομικά βιώσιμες ακριβώς λόγω της καθυστέρησης της αποζημίωσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν εκταμιεύονται αυτά τα ποσά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός ε, Προϋπολογισμός, ο οποίος είναι συγκεκριμένο και για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για τη Γεωργία, είναι είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή ημέρα. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει επάρκεια πόρων για να μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε ή να αναλάβουμε αυτές τις προκλήσεις ε, που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θεωρώ και με αυτό ολοκληρώνω ότι είναι απαραίτητο να εκταμιωθούν αυτές οι ε, ενισχύσεις ε, διότι διακυβεύεται η διαβίωση πολλών μικρών επιχειρήσεων Θεωρώ ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να προέρθει από την Επιτροπή μας, αλλά θεωρώ επίσης και ότι θα πρέπει να είναι κάποιο άλλο ταμείο και όχι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε αυτό που θα πληρώσει τις αμοσμιώσεις αυτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Ριμπέιρο. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι είμαι και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας ε, και έχει γίνει επανειλημμένος αυτή η συζήτηση και εκεί. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι όταν συζητούμε το θέμα του εμπάργου της Ρωσίας θα πρέπει να δούμε και τις συνέπειε τη άμεσης ενισχύση ε, για τις χώρες της Βαλτικές και τις άμεσες συνέπειε για όλες τις χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία υπάρχει άμεση ζημία και ήδη έχουμε και έμεσε ζημίε για το γάλα με μείωση δραστική της τιμής του γάλακτος στην ε, περιοχή μου είχαμε μείωση 2 σέντ το λίτρο ε, για τους γεωργούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2014 ο Επίτροπος Τσόλος ε, ανέλαβε μια σειρά από μέτρα προκειμένου να περιορίσει τις ζημίες και ευπρόσδεκτα αυτά τα μέτρα, αλλά πλέον παρατείνονται τα προβλήματα και η ε, βοήθεια προβλέπεται για ένα χρόνο και τίποτα δεν μας ε, επιτρέπει να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε να κλειτώσουμε τις συνέπειες αυτού του εμπάργου σύντομα. Θα ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε εμπάργο επί εμπάργο επί εμπάργο. Και όσον αφορά το θέμα της επασχόλησης και συζητώντας με την Κομισιόν αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον εγώ αυτό είχα καταλάβει, να μπορέσουμε καταρχήν να δούμε τον αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε εδώ, σε αυτή την Επιτροπή επίσης, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην απασχολησιμότητα ώστε να μπορέσουμε και εμείς εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, να δούμε και να αναλύσουμε τρόπους να καταπολεμήσουμε αυτή τη ζημιά όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Και δυστυχώς αυτό δεν το άκουσα καθόλου στην παρουσίαση της Επιτροπής. Κάποια μελέτη, κάποια εξιολόγηση σε σχέση με τον αντίκτυπο που έχει το εμπάργκο στην απασχολησιμότητα. Και ελπίζω πραγματικά αυτό να γίνει. Η Γεωργία είναι τομέας βασικός στην Ευρώπη και χρειάζεται να δώσουμε αυτή την ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη δημιουργία απασχόλησης χωρίς να δούμε το πρωτογενείς μας τομείς και γι' αυτό είναι σημαντικό ε, η συζήτηση αυτή να γίνει. Και ελπίζω επίσης, σε σχέση με την ανάλυση που έγινε, ώστε να αναζητήσουμε νέες μορφές χρηματοδότησης και επίλυσης του προβλήματος του ρωσικού εμπάργου, πέρα λοιπόν από την αντιμετώπιση των με τον τρόπο που κάνουμε που νομίζω πως είναι τελείως ε, κατάλληλος. Εν πάση περιπτώσει, όταν θα γίνει ε, η συζήτηση για τον προπολογισμό του 2015 να ληφθεί υπόψη ότι οι γεωργοί πρέπει να ε, προστατευθούν γιατί διαφορετικά θα έχουμε ακόμα καλύτερη ανεργία στην Ένωση. Και αυτή η συζήτηση θα γίνεται στην Επιτροπή Γεωργίας γιατί επιβαρύνεται με την παροχή ενός ταμείου αποθεματικού για άλλο στους σκοπούς. Πρέπει να είμαστε συνεπεί. Αν ε, ε, θεωρούμε ότι έχουμε πρόβλημα με το εμπάργκο, το ρωσικό θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα γεωργικά μας προϊόντα απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ. Mr. Thank you very much. ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την ε, Λιθουανία. 20% εξαγωγές στη Ρωσία. Μας επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ το εμπάρκο και το μέσο μεταφορών επηρεάζεται πολύ. Ακόμα μεγαλύτερο είναι εκεί ο αντίκτυπο από τις εξαγωγές της ίδιας των αγροτικών προϊόντων. Έχω μία πρόταση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, για να μην αλλάξει όνομα και να μην ονομαστεί Ευρωπαϊκή εγώ, Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και για το εμπάργκο. Μία λέξη να προσθέσουμε για να μπορεί όποιο θέλει να το χρησιμοποιεί. Πολύ απλά τα πράγματα. Και να ευχαριστήσω την συνάδελφα από την Τσεχική Δημοκρατία που έκανε την πρόταση. Να η λύση. Να η ευκαιρία. Πολύ σοβαρή πρόταση. Μία λέξη να προσθέσουμε και όλοι θα είναι κερδισμένοι. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, να πάνε όλα τόσο εύκολα. Ίσως θα χρειαστεί να προσθέσουμε και λεφτά και όχι μόνο τη λέξη embargo. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ένα πράγμα που είναι ξεκάθαρο ωστόσο είναι ότι όλες αυτές τις ανησυχίες θα τις μεταφέρω στην υπηρεσία μου για να διασφαλίσω ότι θα τροφοδοτηθούν όλα αυτά στις συζητήσεις μας. Ήταν πολύ χρήσιμες λοιπόν αυτές οι παρατηρήσεις, αυτά τα σχόλια, τα κατανόησα πλήρως. Το να προσθέσουμε στο ETF ε, μία λέξη, ξέρετε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα γιατί πρόκειται για ένα νομικό μέσο, για ένα κανονισμό που θα πρέπει να αλλάξει σημαντικά και θα ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός δεν προέρχεται από τον κανονικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά από το παθηματικό. Είναι ειδικό ταμείο, λοιπόν. Και γι' αυτό, λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα και άμεσα. Σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ και τον παγκόσμιο αντίκτυπο, πολύ φοβάμαι ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή τις πληροφορίες που ζητάτε, αλλά σίγουρα θα το μεταφέρω αυτό ω ερώτημα στην υπηρεσία μου. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, συνεργάζονται στενά με τον κλάδο της γεωργίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στις μεμονωμένες χώρες. Ε, Αναφέρατε ότι είσαστε τμήμα, ότι συμμετέχετε στην Επιτροπή Γεωργίας. Αν σας ενδιαφέρει ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, σε ένα λεπτό θα μπορέσει να σας παρουσιάσει το τι γίνεται από δική τους πλευράς. Γιατί πραγματικά ε, συνεργάζονται με την κοινότητα των Γεωργών. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα δώσω το λόγο στους, στον Στη συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια να πω, γιατί πιστεύω ότι τα μέλη της Επιτροπής ε, γνωρίζουν τι γίνεται και γνωρίζετε τι γίνεται στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη σε ό,τι αφορά το εμπάρκο στους παραγωγούς του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες οι οποίες ήδη έχουν αναφερθεί και σε όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε για τις ανισορροπίες της αγοράς που προκλήθηκαν. Υπάρχουν ήδη κάποιες θετικέ τάσεις. Επίσης, πολλά μέτρα ελήφθησαν σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Trade, εμπορίου. για τα φυτογενομικά μέτρα. Υπήρξαν ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι άλλοι συνάδελφοι ε, θα μπορούσαν να σας δώσουν και περαιτέρω πληροφορίες γραπτά αν θέλετε. Αλλά να πω το εξής. Ο, ο Επιτροπός Τσιόλος ξεκίνησε τις κινήσεις για την αποζημίωση της απώλειας εισοδήματος. Είμαστε στη φάση διενέργησης αναλύσεων για το τι θα σήμαινε αυτό συγκεκριμένα. Και φυσικά θα πρέπει μετά την ανάλυση να γίνουν και περαιτέρω συζητήσει γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ κλάδοι. Και ξέρουμε ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι. και κάποια από τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από το ποθηματικό για τις κρίσεις. Ξέρουμε ότι το ποθηματικό αυτό ε, χρηματοδοτείται από τις άμεσες πληρωμές. Είναι δύσκολες λοιπόν οι αποφάσεις ως προς τις πολιτικές κινήσεις, αλλά θα συνεχιστούν σε επίπεδο Συμβουλίου και στην ε, Επιτροπή για τη Γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή θα αρκεστεί στη σημερινή συζήτηση. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Και θα μπει στο θέμα αυτό και σε μελλοντικέ συνεδριάσεις στην ατζέντα. Προσβλέπουμε λοιπόν στις μελλοντικές συζητήσεις τα στις δυνατότητες να αλλάξει το σύστημα γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, ίσως όμως να μπορούν να εξευρεθούν λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν να προσφέρουμε κάτι, έστω περιορισμένο, σε όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Χαιρόμαστε όμως ε, που γνωρίζετε ότι αυτό το θέμα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας όχι μόνο στην Επιτροπή Επασχόληση, όχι μόνο στην Επιτροπή Εμπορίου και στις άλλες αρμόδιες επιτροπές, αλλά και στην Επιτροπή Επασχόληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Και έτσι λοιπόν, αν σωστά κατάλαβα, μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Άλλη μια μελέτη, την οποία και ζητήσαμε. Θέλαμε να γίνει μία μελέτη για την κατανομή των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε πρέον και ο κρύος Κρίστιαν Κέριγκερ, Ενρίκες Λόπες Μπάρτσο, Ράου Δράμος και Βινσέντερ Βαγιέλα και ο κύριος Σορνάκ είναι οι υπεύθυνοι για την μελέτη αυτή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ραούλ Ραμός για να παρουσιάσει την μελέτη. Μία σύντομη εκδοχή της μελέτης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα σας εύχομαι. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας και να σας δώσω το σχετικό feedback. Ήταν ε, μεγάλη και σκληρή η μέρα σήμερα για πολλούς από εσά. Να σας δώσω μια επισκόπηση της μελέτης και ξέρω ότι την είχατε λάβει εκ των προτέρων. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να κάνετε κάποια αρχικά σχόλια, αλλά ασφαλώς και θα είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Να σας παρουσιάσω λοιπόν καταρχάς ε, γιατί ξεκίνησε η όλη ανάλυση. Όπως ξέρετε, η περιξανισότητα τους μισθούς που μας ανησυχούσε από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Αυξήθηκε σε κάποιες χώρες δε. Θα ξέρετε ότι η κρίση επιδίνωσε τουλάχιστον την αντίληψη της ανισότητας στο μυαλό του κόσμου. Άρα, το βασικό ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει η μελέτη είναι τι έγινε με τη μεγάλη ύφεση και πώς επηρεάστηκαν οι τάσεις ανισότητας. Κοιτώντας τα επίσημα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ανισότητα των μισθών, βλέπετε τις πληροφορίες στα μέτρα που χρησιμοποιούν α, τα κρατημέλη για να μετρήσουν τις ανισότητες. των συντελεστή Τζίνι. Κατανομή Το ένα είναι η μέγιστη συγκέντρωση, η μέγιστη ανισότητα. Βλέπετε λοιπόν τι έγινε μεταξύ 2007 και 2011 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίμιση των χωρών αυτών έχουν σημειώσει αύξηση της ανισότητας. Τι κάναμε λοιπόν στη μελέτη αυτή. Συλλέξαμε δεδομένα από επίσημες μελέτες που έγιναν στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντοπίσαμε ποιες ήταν οι τάσεις στην ανισότητα και μετά προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ποιοι παράγοντες επηρέασαν τις τάσεις αυτές. Ένα παράδειγμα. Η ανισότητα δεν αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αν και τα τελευταία δεδομένα που μπορούμε να αναλύσουμε είναι τα στοιχεία του 2011. Δεν ξέρουμε τι έγινε λοιπόν πιο πρόσφατα, το 12, το 13. Έχουμε επίσης ένα οικονομετρικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει κάποια εμπειρικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τους συντελεστές για τις αλλαγές ε, στις τάσεις της ανισότητας. Οι διάφορες οικονομικές δυνάμεις, ε, οι θεσμοί για την αγορά εργασίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο η κρίση. Και επίσης πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες που εξελίχθησαν με άνισο τρόπο. Να κοιτάξουμε τα επίπεδα ανισότητας. Εν συντομία, βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι η κατανομή. Κατά κεφαλή. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διαφορά σε ό,τι αφορά τις, ε, τα ετήσια έσοδα ανά έτος, κατά Βλέπετε λοιπόν τα στοιχεία και παρατηρούμε στην επόμενη διαφάνεια ότι η ανισότητα στο μισθό έχει αυξηθεί κατά δύο, στα δύο τρίτα των κρατών, παρά το γεγονός ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι πολύ σημαντικές. Τι σημαίνει αυτό, ότι η διαφορά μισθών εξηγείται μόνο μέσω των εξελίξεων της ανεργίας και των τάσεων στην αγορά εργασίας και της εξέλιξης των ε, τα συνεργασίας χαμηλού μισθού. Βλέπετε λοιπόν στο αριστερό τμήμα τη διαφάνεια... κάποια αριθμητικά στοιχεία που συγκρίνουν τον μέσο μισθό με το μέσο που λαμβάνουν οι πιο χαμηλόμισθοι. Αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι, το... που είναι κάτω από το 10% του μέσου μισθού. Βλέπουμε ότι στις πιο πολλές χώρες η εξέλιξη ήταν να αυξηθεί αυτός ο αριθμός μεταξύ 2006 και 2011. Και βλέπετε τις χώρες που είναι πάνω από την ε, γραμμή. Στο αριστερό τμήμα βλέπετε τι έγινε στις χαμηλόμιστες θέσεις απασχόλησης. Χαμηλόμιστες είναι αυτές οι θέσεις που λαμβάνουν δύο τρίτα από το σε σχέση με τον μέσο μισθό. Εκεί λοιπόν δεν είναι σαφής η εικόνα από ό,τι βλέπετε. Οι αλλαγές λοιπόν στην ανισότητα κατά την κρίση δεν συνδέονται με τις αλλαγές στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν σε κάποια ε, ιδρύματα που επηρεάζουν την αγορά επηρεάζουν την κατάσταση αυτή. Ένας άλλος στόχος της ε, μελέτης είχε να κάνει με το ρόλο των ε, θεσμικών οργάνων. Κοιτώντας τι έγινε στην κρίση σε σχέση με τρία από τα βασικότερα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τη συλλογική διαπραγμάτευση, το μέσο μισθό και τον ελάχιστο μισθό. Βλέπετε ότι οι ελάχιστοι μισθοί εξελίχθησαν με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που θα αναμενόμε αναμενόταν. Γιατί ο πληθωρισμό στην περίοδο αυτή ήταν υποέλεγχο. Ο ελάχιστο μισθό μειώθηκε σε διάφορες χώρες λόγω προσαρμογής των μισθών κατά την κρίση. Αλλά η αναλογία μεταξύ ελάχιστου μισθού και μέσου μισθού έχει μειωθεί. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των ε, στοιχείων αυτό σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ανισότητας των μισθών. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι ελάχιστοι μισθοί έχουν ε, επηρεάσει την εξέλιξη της ανισότητας, ιδιαίτερα στη χαμηλή, ε, στους χαμηλόμισθους, όπου ο χαμηλή μισθή είναι υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο μισθό, είναι, έχει απαλληλθεί, δεν είναι τόσο μεγάλος ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την ανισότητα. Κοιτώντα τώρα τι γίνεται σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Και αυτό μπορούμε να μοιράσουμε στην έκθεση, δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρεια. Σε ό,τι αφορά την πυκνότητα α, συνδικάτων, σε ό,τι αφορά την κάλυψη από το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές ε, ε, διαπραγματεύσεις, βλέπετε πώς επηρεάζουν το μοντέλο. Κοιτόμαστε λοιπόν, κοιτάμε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη παγκοσμιοποίηση, των τεχνολογικών αλλαγών, των αλλαγών του οικονομικού κύκλου στην περίοδο αυτή και επίση τη οικονομική δομή των διαφόρων χωρών. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι μεγάλο ο τη της παγκοσμιοποίησης τεχνολογικών αλλαγών σε ό,τι αφορά την ανισότητα. Επίση, η βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα επίσης επηρεάζει την, τον ελάχιστο μισθό το τελευταίο τμήμα της μελέτης. Βλέπουμε πόσο είναι καθοριστικοί αυτή οι ε, παράγοντες και εστιάζουμε πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικός είναι ο αντίκτυπος των ημερομυστίων και η εξέλιξη αυτών. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να οφείλονται στην εξέλιξη των μισθών ή των υπόλοιπων ε, πηγών ε, εισοδημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης μπορούμε να διακρίνουμε την εξέλιξη των ε, μισθών, των εισοδημάτων από των ανεξαρτήτων επαγγελματιών, τα εμβάσματα ή άλλα εισοδήματα, καθώς και την, τον αντίκτυπο των φόρων, της φορολόγησης. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, ανάμεσα στο 2006 και το 2011, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι ανισότητα των μισθών φυσικά οδηγεί στην ανισότητα των εισοδημάτων και επηρεάζει τη συνοχή στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι δηλαδή θετικό και Όσο η μεγαλύτερη είναι η ανισότητα των μισθών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανισότητα των εισοδημάτων. Ε, ε, και επηρεάζεται και οι αλλαγές στην ανισότητα όσον αφορά τις διάφορες πηγές ε, εισοδημάτων. Τα επιδόματα αλλά και οι φόροι, αν είναι σωστά σχεδιασμένα, θα πρέπει να μειώσουν την απόλυτη ανισότητα. Και αυτό το βρίσκουμε περισσότερο στους φόρους, αλλά όχι τόσο σε θέματα επιδομάτων. Τελικό, ένα βασικό συμπέρασμα μάλλον είναι ότι η ανισότητα, ανισότητα των μισθών ε, ε, παίζει ρόλο στην ανισότητα των εισοδημάτων, αλλά δεν είναι ο κύριος παράγοντας. Υπάρχουν και κάποιες οικονομικές ε, πηγές που εξηγούν την ανισότητα της εξέλιξης. Ευχαριστώ πολύ. The floor is open. We can put questions. Μπορείτε τώρα να θέσετε ερωτήσεις αν το επιθυμείτε. Ιούτα viel... Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Είναι πάρα πολύ κρίμα που η μελέτη φτάνει μόνο μέχρι το 2011. Γιατί μετά το 2011 είχε ενδιαφέρον και σίγουρα τότε υπήρξαν οι μεγάλες επιπτώσεις. Λέτε ότι δεν αυξήθηκαν οι ανισότητες. Εγώ φαντάζομαι ότι τα τελευταία τρία χρόνια με την πολιτική λιτότητα. Η κατάσταση αυτή θα έχει αλλάξει. Αν ε, μου επιτρέπετε να συνοψίσω τα ε, συμπεράσματα, μειώθηκε μειώθηκαν οι μισθοί στο σύνολό τους με την κρίση. Αυτό είναι φυσικά αρνητικό και για την οικονομία και οι πολιτικοί λιτότητες επιδίνωσαν την κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη. Είπατε ότι ο πιο μεγάλος ανταγωνισμός, η πιο μεγάλη απορρίθμιση θα είχε τεράστιο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τις ανισότητες, τις μισθολογικές. Έχετε κάποιους συγκεκριμένους τομείς να μας δώσετε ως παραδείγματα. Και να μας πείτε πώς επιδεινώθηκε το θέμα της ανισότητας των μισθών. Κοιτώντας την οικονομία στην Ευρώπη και τα προϊόντα που παράγονται. Πώς μπορεί να δοθεί κίνητρο στην ιστορική ζήτηση. Ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. και μέσω της μείωσης των μισθών δεν προκύπτει και μείωση των φορολογικών εισόδων. Μείωση των εισφορών στα κοινωνικά συστήματα, στα συνταξιωτικά συστήματα. Πώς επιτράει ο παράγοντας αυτός. Τελευταίο σημείο. Αν κατάλαβα σωστά, οι συλλογικέ συμβάσεις των κοινωνικών εταίρων δεν είναι πλέον δεσμευτικοί. Και όσο πιο, δεν είναι, όσο πιο πολύ δεν είναι δεσμευτικέ οι συλλογικέ συμβάσει, τόσο μεγαλύτερε είναι οι ανισότητε. Άρα, όντω, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συλλογική αυτονομία για τι ε, συλλογικέ συμβάσει. Όπω υπήρχε σε κάποιες χώρες, θα πρέπει να επανέλθουμε στο μοντέλο αυτό. Okay, for, Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και το σχολείο σας. Συμφωνώ ότι είναι κρίμα που δεν μπορούμε να εξετάσουμε πιο πρόσφατα στοιχεία για αυτή τη μελέτη, αλλά αυτό δεν είναι μέσα στο πεδίο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα για τα εισοδήματα ε, και τις συνθήκες διαβίωσης είναι εξάλλου αυτό απαραίτητο γιατί είναι μια μεγάλη στατιστική επιχείρηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε λοιπόν. Τώρα, σε σχέση με τον αντίκτυπο της ανισότητας των, ε, των μισθών όσον αφορά την έξοδο από την κρίση και πώς ε, η απώλεια αγοραστικής δύναμης έχει επηρεάσει ή επηρεάζει την ανάκαμψη κάποιων κρατών μέλων, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Η ανισότητα ειμαστε απολυτα συμφωνοι η ανισοτητα μισθων είναι πολύ πιο ε, έντονη στο χαμηλότερο τμήμα των μισθών και αυτό επηρεάζει ε, τους φτωχότερους εργαζόμενους στις διάφορες χώρες και αυτό είναι αυτό που επηρεάζει την κατανάλωση, τη ζήτηση και ούτω καθεξής. Ε, ακόμα και αν λάβουμε υπόψη λοιπόν τον αντίκτυπο στον μέσο άνθρωπο, σε κάποιες ε, χώρες ε, ο πληθωρισμός των μισθών έχει συνοδευτεί από ψηλότερη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές, οπότε βοήθησε στην απόδοση την εξαγωγική των λόγων χωρών, είναι δηλαδή πιο δύσκολο να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει μόνο εξετάζοντας τον αντίκτυπο στην κατανάλωση. Πάντως αυτό ήταν ένας από τους στόχους του προγράμματος που είχε, όχι, ήταν, δεν ήταν αυτός ο στόχος του προγράμματος, ήταν να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και όχι ποιες είναι οι συνέπειες. Αλλά θα ήταν και αυτό πολύ ενδιαφέρον να, να μελετηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Εάν όχι, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε και το είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί όταν θα σας αναθέσουμε την επόμενη έκθεση σε ένα-δύο χρόνια θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε την κατάσταση που θα ισχύει μετά την κρίση. Νομίζω λοιπόν πως όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι πολύ χρήσιμες και για την Γιούτα Στάινρουκ και για μένα. Και για άλλους που συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή και που επιθυμούν να